Proszę Państwa, z pewnym opóźnieniem, ale jak Państwo zauważyli... Καλημέρα σας. Έχουμε λίγο καθυστερήσει, αλλά όπως τα είδατε, έχουμε και ένα προσκεκλημένο. Τον Επίτροπο. Μάλιστα ήρθε και πρώτος. Μας πρόλαβε, μετά ήρθαμε εμείς. Και χρειάστηκε να περιμένουμε μέχρι να γεμίσει κάπως η αίθουσα για να αρχίσουμε τις εργασίες μας. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Σας καλωσορίζω με αυτή την αιαρινή άβρα. Ξέρετε ότι η άνοιξη έχει μεγάλη σημασία για τους γεωργούς, για τις γεωργικές εργασίες. Ελπίζω να είναι πρόσφορο και για τις εργασίες της δικές μας. Καλώς ήρθατε. Αρχίζουμε με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας, των πρακτικών της ως 23 και 24 Φεβρουαρίου. Στις ανακοινώσεις του Προέδρου έχω να σας πω μόνο ότι έχουμε τις συνήθεις γλώσσες 20 δηλαδή πλην εσθονικών, μαλτέζικων, σλοβακικών και ιρλανδικών. Ξεκινώ με τον Επίτροπο, τον οποίο και καλωσορίζω, τον κύριο Άντριου Κάιτης υπεύθυνο για την υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων, που έρχεται για πρώτη φορά στην Επιτροπή μας να μιλήσει για θέματα ασφάλειας τροφίμων. Έχουμε πολλά σημαντικά θέματα που συζητούμε εδώ στην Επιτροπή μας. Θέματα αρμοδιότητάς του, θέματα που απασχολούν και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια σειρά από προβλήματα που θα δούμε και στην ημερήσια μας διάταξη στο σημείο 5. Το βακτηρίδιο κλεψιέλα που πλήττει τις, τα ελαιόμετρα της Ευρωπαϊκής Μεσογείου και άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Για άλλη μια φορά λοιπόν ευχαριστώ και καλωσορίζω τον Επίτροπο και τους συναδέλφους που τον συνοδεύουν. Χωρίς να καθυστερούμε λοιπόν άλλο, σας δίνω το λόγο κύριε Επίτροπε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν ήθελα να σας καθυστερήσω. Έχω μόνο ένα αίτημα γιατί ήθελα να ζητήσω την αλλαγή της ημερήσιας διάταξης. Να καταθέσω τώρα το αίτημα ή να περιμένω πρώτα να ακούσουμε τον Επίτροπο και μετά να κάνουμε τη συζήτηση αυτή. Δεν θέλω να σας καθυστερήσω άλλο. Μπορούμε να το κάνουμε και μετά. E, Κοιτάξτε, κανονικά αυτά είναι τα θέματα που συζητούμε στην αρχή, αλλά αν θέλετε μπορείτε να τοποθετείτε μετά τον Επίτροπο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας και που έχω την ευκαιρία να συζητήσουμε μια σειρά από θέματα που μας ενδιαφέρουν όλους από την άποψη της ασφάλειας των τροφίμων. Εδώ και πέντε μήνες ανέλαβε η νέα Επιτροπή τα καθήκοντά της και έκτοτε έχω κοιτάξει τις καταθυντήριες γραμμές που έχει δώσει ο πρόεδρος Γιούγκερτ και τις έχω συνδέσει με την επιστολή αρμοδιοτήτων μου. Έχω κοιτάξει τι έχει γίνει από την ε, πρώην Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ σε σχέση με την εντολή που αναλαμβάνω. Και εγώ με τι υπηρεσίε μου και του συνεργάτε μου έχουμε ετοιμάσει μια σειρά από προτεραιότητε για του δύο βασικού ε, πυλώνε πολιτική. Την υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων για το 2014-2019. Σκοπεύουμε να έχουμε μια σφαιρική προσέγγιση και για του δύο πυλώνε και ένα όραμα για την ερχόμενη πενταετία. Ελπίζω ότι στο μέλλον θα είμαστε σε θέση να έχουμε συστηματική ενημέρωση για την κατάσταση τη υγεία στην Ευρώπη και ιδιαίτερη ε, προσοχή στην ε, ασφάλεια των τροφίμων καθώς και τις σχετικές πολιτικές σε όλα τα κράτη-μέλη. Ελπίζουμε ότι έτσι θα βελτιστοποιήσουμε την προστιθέμενη αξία της ευρωπαϊκής ε, προσπάθειας. Παράλληλα, έχω φροντίσει να συναντηθώ επανειλημμένως με τους συναδέλφους επιτρόπους, με μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων, υπουργούς και άλλους ενδιαφερομένους, με κυβερνητικές οργανώσεις, εκπροσώπους των εταιριών, την κοινωνία των πολιτών και είχαμε επικοδομητικές ε, συζητήσεις. Βεβαίως κάποιες παρουσίασαν δυσχέρειες για τα θέματα που συζητήσαμε, αλλά αυτό είναι κάτι που ε, εντάσσεται στα πλαίσια της όλης προσπάθειας. Ε, άκουσα προσεκτικά ό,τι είχαν να πούν οι συνομιλητές μας, αλλά αυτές οι ανταλλαγές ήταν πραγματικά μια ευκαιρία να σφιγμομετρήσουμε την πραγματικότητα. Σήμερα θέλω να σας δώσω μια ευρύτερη εικόνα του πυλώνα για τα τρόφιμα που αυτή τη στιγμή περατώνουμε εσωτερικό στις υπηρεσίες της Επιτροπής. Πριν ξεκινήσω όμως να πάω σε κάτι που ενδιαφέρει όλους, ιδίως εσάς τους πολιτικούς, γιατί Απρόκειται για την ανάπτυξη και τι θέσει εργασία. Θα πρέπει εδώ να ε, συνεργαστούμε βάσει των συνθήκων και να επισημάνω την προσοχή σα στο άρθρο 168 τη συνθήκη για τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να φροντίσουμε το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή να εντείνουν τη συνεργασία του με τα κράτη-μέλη, ώστε να υπάρχει ενό υψηλού επίπεδου προστασία τη ανθρωπίνη υγεία με σωστού ορισμού και υλοποίηση όλων των πολιτικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών δράσεών τη. Αυτό είναι το δικό μα μερίδιο Βεβαίω, Έχουμε και ο καθένα τι προτεραιότητέ του. Ε, εγώ βάσει των προτεραιοτήτων που ορίζονται και από την επιστολή του, Ιου, του κυρίου Γιούνκερ, εσεί βάσει τη αποστολή που αναλάβατε εκλεγόμενοι και ω πρώην μέλο ε, του Κοινοβουλίου για περισσότερα από 20 χρόνια, πρέπει να πω ότι σέβομαι την εντολή σα ε, που προέρχεται από του ίδιου του ψηφοφόρου. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου βεβαίω ότι όλοι υπηρετούμε του Ευρωπαίου πολίτε. Είμαστε εδώ για να βεβαιωθούμε ότι σε πέντε χρόνια οι άνθρωποι θα ζήσουν, θα καταλάβουν τη διαφορά από τι πολιτικέ μα, ώστε μέχρι τι επόμενε εκλογέ να μην δείξουμε απλώς ότι κάναμε θετικές αλλαγές, αλλά ότι ε, δεν χρειαζόμαστε να φοβόμαστε ότι θα υπάρξουν ακραίες τάσεις. Να σας πω τώρα ποιες είναι οι δικές μου προτεραιότητες. Ε, επί της ουσίας νομίζω ότι καλύπτουν τις ανάγκες των δικών σας ψηφοφόρων ε, με τον ίδιο τρόπο που και εσείς θα θέλατε. Υπάρχουν νομοθετικές προτάσεις για τις οποίες θα σχολιάσω αργότερα, αλλά οι προτεραιότητες που έχω εντοπίσει εγώ στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων καλύπτουν την διαχείριση των κρίσεων, την επισητιστική ασφάλεια και τη βελτίωση της νομοθεσίας, την αναθεώρηση της ε, διαδικασίας λήψης αποφάσεων για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς και τους ενδοκρινικούς ε, διαταράκτες και την ε, αντιβιωτική αντίσταση, την αντιμικροβιωτική αντίσταση, την ασφάλεια των τροφίμων και την υγεία των ζώων. Εδώ να σταθώ σε καθένα από αυτά τα θέματα. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την ε, πρώτη αποστολή που ανέλαβα από τον πρόεδρο Γιούνκερ, την πρώτη υποχρέωση, διότι πρέπει ο κάθε επίτροπος να διδραματίζει το ρόλο του στην στήριξη των δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην αντιμετώπιση κρίσεων. Βλέπετε την κατάσταση με τον ε, πυρετό των ε, χείρων, με την γρήπη των χείρων και το σχετικό κρούσμα. Το πρώτο που ανέλαβα είναι να βεβαιωθούμε ότι η κατάσταση θα παραμείνει εντό ελέγχου και ότι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση σε αυτή την περιοχή. Αυτή είναι η καθημερινή μου δουλειά. Η δεύτερη αρμοδιότητά μου είναι να εξυγχρονίσω και να πλουστεύσω την ισχύωση νομοθεσία. Επ' αυτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να μειώσει το γραφειοκρατικό άχθο στι όλε διαδικασίε και δράσει που προβλέπονται για τι εταιρείε τροφίμων και του σχετικού φορεί. Η τρίτη πτυχή είναι εδώ τον, η πτυχή των εισαγωγών των μη συμμορφωμένων προϊόντων με την νομοθεσία μας. Εδώ επηρεάστηκαν όλοι οι τομείς των επενδύσεων και η βιομηχανία των τροφίμων κατά κύριο λόγο. Είμαι αποφασισμένος να αντιμετωπίσω αυτούς που δεν σέβονται τους κανόνες μας και να ε, ε, αναλάβω όλες τις σχετικές δράσεις. Όταν ολοκληρώσουμε την αναθεώρηση των κανόνων για τους ε, ανεπίσημους ελέγχους, σκοπεύω να ασχοληθώ ε, ιδιαίτερα με το θέμα των μη συμμορφούμενων ή μη ασφαλών προϊόντων, ιδίως όσων ε, προέρχονται από τρίτες χώρες. Για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις αθέμητες πρακτικές πρέπει να έχουμε και τη στήριξη των υπολείπων αρχών, όπως των τελωνιακών, των φορολογικών και όλων των υπολείπων. Τώρα να στραφώ στα γενετικώς τροποποιημένα. Όπως ε, θα γνωρίζετε, καταφέραμε να συμφωνήσουμε την συνέχεια που θα δώσουμε στην πολιτική αυτή. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ξανά όλους στο Κοινοβούλιο γιατί δείξατε ότι ακόμα και σε ευάλωτα και δυσχερή ζητήματα, ε, σε ευαίσθητα μάλλον και δυσχερή ζητήματα, μπορείτε να έχετε φιλόδοξες προτεραιότητες και να προτείνετε σωστές λύσεις. Ε, η κοινή μας πρόκληση, βάσει και των όσων ε, έχει ορίσει ο πρόεδρος Γιούνκερ, είναι να θεωρήσουμε τη διαδικασία έγκρισης για τους γάμματα φόμικρον και τα προϊόντα, τα σχετικά προϊόντα. Υπό αυτήν την έννοια, η διαδικασία λήψης αποφάσεων ε, δεν έχει ακόμη περατωθεί. Θα ολοκληρωθεί και θα δημοσιευτεί στο τέλος του Απριλίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επανειλημμένω έχει κληθεί να ανταποκριθεί στι προσδοκίε των πολιτών και πραγματικά ανυπομονώ να έχουμε οικοδομητικό διάλογο μαζί σα αλλά και εν τέλει να βρούμε τις λύσεις που χρειαζόμαστε για να αναλάβουμε τις ευθύνες μας ως ε, ε, εκλεγμένοι δημοκρατικά. Ε, εσείς δηλαδή και εμείς ως Επιτροπή. Τώρα για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Πριν από δύο εβδομάδες ψηφίσατε για το θέμα αυτό στην Ολομέλεια. Δεν θα αναπτύξω πλήρως το θέμα αυτό στις λεπτομέρειες του, απλώς να επαναλάβω τη δέσμευσή μου, να αναλάβω ταχεία δράση με συνθήκες πλήρους διαφάνειας και να ικανοποιήσω τις ε, ανάγκες των πολιτών κατά πρώτο λόγο. Ε, εδώ ελπίζουμε ότι θα συνεχίσετε κι εσείς να ευαισθητοποιήσετε για το θέμα αυτό και να ευαισθητοποιείτε τους υπολείπους και θα συμμετέχετε στις συζητήσεις που προγραμματίζω να οργανώσω για τα ενδιαφερόμενα μέλη του Κοινοβουλίου στις 23 Απριλίου και στη δημόσια διάσκεψη που θα οργανωθεί αργότερα. Ε, ένα άλλο σοβαρό θέμα, κατά την άποψή μου, είναι η αντιμικροβιακή αντίσταση. εδώ πρέπει να διαφυλάξουμε την δράση των αντιβιωτικών. Είναι ένα σημαντικό ε, στοιχείο που διαθέτουμε για να καταπολεμήσουμε νόσους και ασθένειες. Εδώ πρέπει να είμαστε βέβαιοι για την δραστικότητα αυτών των αγωγών, διότι ε, μειώνεται όταν δεν χρησιμοποιούνται σωστά. Έτσι, Το AMR έχει γίνει, η αντιμικροβιακή δηλαδή αντίσταση, έχει γίνει μια από τις πρώτες μου προτεραιότητες ε, και η αντιμετώπιση της. Το έχουμε συζητήσει ήδη στο Κοινοβούλιο και έχουμε αντιμετωπίσει το θέμα στο πλαίσιο των φαρμακευτικών ζωοτροφών αλλά και των κτηνιατρικών φαρμάκων. Εδώ λοιπόν σε ό,τι αφορά τι φαρμακευτικέ ε, ζωοτροφές χαίρομαι που ήδη προτείνονται μέτρα για να καταπολεμήσουμε την αντιμικροβιακή αντίσταση ιδίω για τι ε, απαγορεύσει για, ε, για συγκεκριμένες συνταγές για ιού και λοιμώξει. Εδώ υπάρχει ισχυρή στήριξη. Θέλω να συνεχιστεί το πρόγραμμα δράση που ήδη εφαρμόζεται και επειδή εκπνέει το 2016 να προβλέψουμε τη συνέχιση του. Επίσης θα πρέπει να προβλέψουμε μέτρα για να συνεχίσουμε την όλη προσπάθεια και θα παραμείνω πιστός στην, υποχρέ... στην δέσμευση που ανέλαβα να συνεχιστεί ο διάλογός μας και να έχουμε μια υψηλή επίπεδου διάσκεψη για το θέμα αυτό προκειμένου να αποτιμήσουμε τι περαιτέρω δράσεις μπορούν να διασφαλίσουν μια καλή συνέχεια. Σε ό,τι αφορά την υγεία των ζώων, η ισχύουσα στρατηγική για την υγεία των ζώων θα ολοκληρωθεί φέτος. Πολλά έχουμε πετύχει και στον τομέα αυτό. Η Ένωση συνολικά με το μοντέλο που έχει καθορίσει για την υγεία των ζώων και τα πρότυπά του έχει καταφέρει πολλά. Όμως υπάρχουν και άλλα σημαντικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, ιδίως ως προς την υλοποίηση. Οι, ε, οι υπόλοιπε επιλογέ πρέπει να μελετηθούν, όπω την ανανέωση τη στρατηγική για να προτείνουμε ένα νέο πρόγραμμα δράση, να, βελτιώσουμε τη χρήση της, ε, την αξιοποίηση τη αρχή τη επικουρικότητα και να δούμε την ημερομηνία εκπνοή τη στρατηγική για την υγεία των ζώων, ώστε να προβλέψουμε τα επόμενα βήματα. Είμαι βέβαιος όμως ότι και εσείς θα συμφωνείτε. Πριν προχωρήσω πρέπει να δούμε το ευαίσθητο αυτό ζήτημα ε, μαζί με τους ε, συναδέλφους μου στο Σώμα των Επιτρόπων. Επίσης, να προσθέσω λίγα λόγια για για τα απόβλητα τροφίμων. Εδώ πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτό είναι ένα θέμα που έχει υψηλή προτεραιότητα στην παγκόσμια ατζέντα για το μέλλον των τροφίμων και της παραγωγής τροφίμων και θα συζητηθεί πολύ σύντομα στη σχετική διάσκεψη σε λιγότερο από έξι εβδομάδε. Εδώ σκεφτόμαστε το τι μέλλον θα έχει αυτή η πολιτική, πώ θα πρέπει να εξελιχθεί και ε, πώ θα προχωρήσουμε και στα πλαίσια τη κυκλική οικονομία. Τελευταίο και όχι λιγότερο σημαντικό, λίγα λόγια για την επισήμανση των τροφίμων. το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την προέλευση των τροφίμων και για την ε, διάσταση που έχουν πάρει άλλα θέματα, όπως κλωνοποίηση τα τελευταία χρόνια. Το Κοινοβούλιο έχει προβλήψει υποχρεωτική επισήμανση ε, για το επεξεργασμένο κρέας ε, και τα προϊόντα του, αλλά βάσει των μελετών μας οι καταναλωτές δεν θέλουν να επομιστούν το επιπλέον κόστος για τέτοιου είδους πληροφόρηση. Έτσι, δεν είμαι ακόμη πλήρως πεπισμένο σε ποιο βαθμό θα έπρεπε ή θα μπορούσε να επιβληθεί υποχρεωτική επισήμανση για το ευρωπαϊκό επίπεδο τουλάχιστον. Πρόεδρε, Κυρίε και κύριοι βουλευτές, επιτρέψτε μου να πω λίγα λόγια για, από για ορισμένα από τα θέματα που μας απασχολούν τώρα και περνούν από την νομοθετική διαδικασία αυτόν τον καιρό. Να ξεκινήσω με την πρόταση για την υγεία των ζώων. Εδώ ε, είμαι ικανοποιημένο με την πρόοδο που έχει τελεστεί ω τώρα στου διαλόγου μα και θέλω να σα ευχαριστήσω, Πρόεδρε, ε, και εσά και του συναδέλφου σα, αλλά ιδίω ε, την εισηγήτρια, την κυρία Πάλσεν, για την επικοδομητική του στάση, για την επικοδομητική σα στάση και τι προσπάθειε να βρούμε από κοινού μια λύση. Με την πρόταση αυτή προσπαθούμε να βελτιώσουμε τα πρότυπα της υγείας των ζώων και να προσφέρουμε ένα πλουστευμένο σύστημα για να ανοιχνεύουμε και να ελέγχουμε τις μεταδιδόμενες νόσους των ζώων. Εδώ να προσθέσω ότι η πρόταση αυτή σκοπό δεν έχει να ρυθμίσει τις κτηνιατρικές ε, ε, αντιμετωπίσεις της υγείας των ζώων. Αυτό θα το δούμε στο ανάλογο νομοθετικό πλαίσιο. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έναν κανονισμό για τις ζωοτεχνικές διαδικασίες σκοπεύει να προάγει το ελεύθερο εμπόριο στην αναπορογή των ζώων, το, την εμπορία και τα τελικά προϊόντα, βεβαιωνόμενοι ότι υπάρχουν βιώσιμα προγράμματα αναπαραγωγής και η προστασία των γενετικών πόρων μας. Να συγχαρώ τον εισηγητή, τον κύριο Νταντάν, ο οποίος ε, είχε επιτυχή δικαιολογημένη και ε, σωστή στάση για την παράταση της πρότασης αυτής. Ε, το συζητήσαμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντο του Κοινοβουλίου το θέμα αυτό. Πρέπει όμω να σκεφτούμε προσεκτικά εάν το δικαίωμα εγκατάσταση και παροχή υπηρεσιών ε, των εταιριών θα πρέπει να περιοριστεί ενδεχομένω για λόγου διαφορετικού πέραν τη προστασία τη ε, βιοπικιλότητα. Τώρα, για την υγεία των φυτών, η Επιτροπή πρότεινε την ενίσχυση των προστατευτικών μέτρων κατά των ε, ε, νόσων των φυτών. Θα πρέπει εδώ να αντιμετωπίσει και να ασχοληθεί και το Κοινοβούλιο Συμβούλιο πολύ σοβαρά με το θέμα αυτό για να βρούμε μια συμβαστική πρόταση μαζί με το Συμβούλιο στους επερχόμενους τριμερείς διαλόγους. Για το θέμα της υγείας των φυτών πιστεύω ότι θα, είσαστε, θα έχετε επίγνωση της ε, πολύ σοβαρής κατάστασης που έχει προκαλέσει η κλεψιέλα. Ε, μια, ένα νέο βακτηρίδιο που επηρεάζει τον ε, παραγωγή ελαιόλαδου στην περιοχή της Απουλίας, στα νότια της Ιταλίας. Οι εμπειρογνώμονες επισημαίνουν ότι 10% όλων των ελαιόδεντρων στην περιοχή αυτή έχουν πληγεί. Και εκεί ξέρουμε ότι η γεωργία εξαρτάται από την παραγωγή ελαιόλαβου. αυτή η νόσος λοιπόν είναι καταστροφική στις συνεπίες της. Επιπλέον οι επιστήμονες έχουν καταλήξει πρόσφατα στο συμπέρασμα ότι τα σταφύλια, τα κλίματα και οι λεμονιές, ε, τα εσπεριδοειδή μπορούν να γίνουν φορεί τη ασθένεια αυτή. Πρέπει να λάβουμε λοιπόν γεωργικά μέτρα στι περιοχέ αυτέ και να προβλέψουμε, να καταπολεμήσουμε την εξάπλωση του βακτηριδίου. Αυτή τη στιγμή ελέγχουμε την κατάσταση και έχουμε ενθαρρυντικά στοιχεία για την ε, πολιτική προφύλαξη που έχει ήδη σχεδιαστεί για την ε, ε, αντιμετώπιση τη εξάπλωση αυτή τη ασθένεια και προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο. Πρόκειται να πάω στην Ιταλία και να επισκεφτώ την πληγήσα περιοχή του Λέτσε γιατί είναι σημαντικό όσοι έχουν ζημιωθεί από αυτό το βατρίδιο να δουν τη δέσμευση της Ένωσης να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Να προσθέσω ότι παρόμοια ε, προσοχή θα δώσω στους παθογενείς παραγόντες στα τρόφιμα. Τα ανησυχητικά επεισόδια του καβυλοβακτηριδίου και της αλμονέλας πρέπει να αντιμετωπιστούν. Έχουμε περίπου 200.000 κρούσματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πέρσι σε ανθρώπους και το 80% των ε, σπαγίων των πουλερικών έχουν ε, μολυνθεί. Πρέπει λοιπόν να αποφύγουμε κάθε περίπτωση να διωγγωθεί ο αριθμό των κρουσμάτων. Είναι ανησυχητικό αυτό που συμβαίνει και πρέπει να το δούμε και στι δημαρει ε, συναντήσει ε, μαζί σα. Τελευταίο και όχι λιγότερο σημαντικό να αναφέρω πολύ σύντομα και την ε, όλη συζήτηση κατά τις διαπραγματεύσεις για το TTIP, την ε, Διατλαντική Εταιρική Σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών. Ε, για τα πρότυπα της ασφάλειας των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα συζητήσουμε θέματα τέτοια, γιατί υπάρχει υψηλό επίπεδο ομάδα για να ασχοληθεί ακριβώς με αυτά. Θα πρέπει να είμαστε σταθεροί στις απόψεις μας και στις σχετικές συνομιλίες με τη Ρωσία για να δούμε κατά πόσο μπορεί να ξανανοίξουν οι εξαγωγές τροφίμων. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να αποδεχτούμε καταστάσεις όπου οι διαφορετικές, διαφορετικά μέτρα και σταθμά να ισχύουν για τα διαφορετικά κράτη-μέλη. Θα πρέπει στα υγειοφυτονομικά ε, μέτρα να δούμε εάν οι εξαγωγές από τη Ρωσία ε, αυξάνονται. Γιατί παρά τις επιτυχίες μας στον περιοχή περιορισμό της γεωγραφικής εξάπλωσης της Αφρικανικής Πανόλης των Χείρων, η Ρωσία διατηρεί δυσανάλογη στάση ε, στους ζώντες χείρους ε, και τις εξαγωγές τους από και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Επιτροπή έχει ξεκινήσει μια διαδικασία επίλυσης διαφοράς ε, μεταξύ Ρωσίας στο επίπεδο του ΠΟΕ για το τόσο ευαίσθητο αυτό θέμα ε, και προκειμένου να προασπιστεί συνολικά τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σας διαβεβαιώσω ότι μόνον εάν η Ρωσία Ρωσία σεβαστεί τη Διεθνή Αρχή της Περιφερειοποίησης ως, ε, ως προς την, μεγάλη, την, παραγωγή μεγάλων, την, την παραγωγή εμπορικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο τότε θα μπορέσει να βρεθεί λύση. Ε, η, Πολλά είναι τα κράτη που έχουν ε, πληγεί από αυτή την απαγόρευση και συνεργάζομαι στενά με τον Επιτροπο Χόγκαν για να βρούμε ποια είναι τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει να αναλυφθούν. Επίση, υπάρχουν ε, και άλλοι επίτροποι που θα συνεργαστούν μαζί μα για να δούμε το άνοιγμα των αγορών στι νότιε χώρε, γιατί για τον ένα ή τον άλλο λόγο υπάρχουν αυτή τη στιγμή δυσκολίε και πάυσει στι ε, εξαγωγέ μα και χρειάζεται μια όθηση σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο. Πρόεδρε, πρέπει να πω ότι τη θέση μου την έχω ήδη περιγράψει σε μια σειρά από θέματα για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε και εσείς και η Επιτροπή σας το τι συμβαίνει. Πρόκειται να διασφαλίσω υψηλά πρότυπα ασφάλεια των τροφίμων για τους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτός είναι ο στόχος μου και θα πρέπει να κινηθούμε από κοινού μπροστά για όλα αυτά τα ζητήματα. Η επιτυχία μας εξαρτάται από το κατά πόσο η προσπάθειά μας θα είναι κοινή. Μόνο έτσι θα έχουμε θετικά αποτελέσματα και θα συνεχιστεί η προσπάθειά μας ώστε σε πέντε χρόνια να βρεθούμε πάλι εδώ και να πούμε ότι δεν θέλαμε απλώς να τα καταφέρουμε αλλά ότι όντως τα καταφέραμε. Ελπίζω ειλικρινώς ότι παρόλο που μπορεί να αντιμετωπίσουμε δυσκολίες, παρόλο που μπορεί να έχουμε και κάποιες διαφωνίες, παρόλα αυτά θα καταφέρουμε να συνεργαστούμε ε, σε ε, ένα πνεύμα θετικό για προς όφελος των πολιτών μας. Τώρα με τα χαράς να ακούσω τις απόψεις σας για όλα αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Πράγματι παρουσιάσατε ένα μεγάλο αριθμό θεμάτων και προβλημάτων με τα οποία καλούμεθα να παλέψουμε. Αυτό όμως και περιμέναμε από πλευρά σας. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι που έχουν ζητήσει το λόγο. Αναφερθήκατε όπως είπα σε πολλά και διαφορετικά θέματα. Θα ακολουθήσουμε την εξής αρχή. Λοιπόν, δύο λεπτά για τους συντονιστές, ένα λεπτό για τα μέλη. Θα σας παρακαλέσω να μην επαναλαμβάνετε αυτά που λένε άλλοι συνάδελφοι, έτσι ώστε να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Ο κύριος Ντες έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, κύριε Ανδρικάητης που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Ναι και δεν έχω πολύ χρόνο, θα περιοριστώ σε ένα σημείο. Την μικροβιακή αντοχή ή αντοχή στα αντιμικροβιακά. Έχετε βέβαια τα θέματα της ασφάλειας των τροφίμων, της ε, υγείας των ζώων και γνωρίζετε πολύ καλά πόσο σημαντικά είναι αυτά για την Ευρώπη. Έχουμε ένα σύστημα ποιοτικό μικροβιακής παρακολούθησης της αντιμικροβιακής ε, ε, αντοχής. Καταγράφουμε το κάθε τι και μπορούμε να καταλήξουμε στη Γερμανία στα συμπεράσματα τα σχετικά με την ε, μικροβιακή αντοχή και τις αιτίες τους. Πρόκειται για ένα σύστημα μοναδικό, το οποίο δεν υπάρχει όμως αντίστοιχα για την υγεία του ανθρώπου, για τη δημόσια υγεία. Μήπως λοιπόν πρέπει να κοιτάξουμε και αυτή την προσέγγιση, ώστε να καταγράφεται και να τεκμηριώνεται το φαινόμενο αυτό και από πλευρά της υγείας του ανθρώπου. Γιατί έχουμε πάρα πολλά αντιβιωτικά όπως ξέρουμε, ε, τον οποίων μικρό ποσοστό μόνο χρησιμοποιείται στα ανώ, έχουμε αντίστοιχα 47% ποσοστό των διαθέσιμων αντιβιωτικών που χρησιμοποιείται τακτικά στον άνθρωπο. Πρέπει και εκεί λοιπόν να γίνει σχετική έρευνα. Επίσης κύριε Επίτροπε χαίρομαι που είπατε ότι σκοπεύετε να αναπτύξετε αγαστή συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Σας έχω γνωρίσει και προσωπικά και ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος με πολλές γνώσεις, με πολύ καλές προθέσεις. Ελπίζω λοιπόν ότι θα έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία στην επόμενη πενταετία με Και αυτό το λέω εκ μέρους και ολόκληρης της ομάδας. Με ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κύριος Μπερέγκα. Ρεμπέγκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξ ονόματος του κυρίου Ντεκάστρο θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να επιβάλλει την εκρίζωση των μολυσμένων ελαιοδένδρων. Και μιας και υπάρχει και μία απαγόρευση ε, να φυτευθούν νέα ελαιόδενδρα, τότε καταλαβαίνετε ότι σε ορισμένες περιοχές ένα τέτοιο μέτρο δεν μπορεί να λειτουργήσει. Υπάρχει επίσης επιμόλυνση και σε γειτονικές περιοχές. Η κατάσταση στον τομέα αυτό, ε, τον φυτολογικό, είναι πάρα πολύ σοβαρή και υπάρχει και πρόβλημα σε σχέση με τις μετασφορές. Κατανοώ την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκρίζωση των ελαιοδένδρων, λαμβανωμένων υπόψη όμως των απολειών που έχουν ήδη σημειωθεί και αναφέρομαι την οικονομική ζημιά των παραγωγών, λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό της επιμόλυνσης και λαμβάνοντας υπόψη ότι το βακτήριο αυτό προέρχεται από την Κοσταρίκα. Ε, έχει δημιουργηθεί μια παράδεκτη κατάσταση. Ε, υπάρχει μια τεράστια περιφέρεια που έχει θυγεί, οι οικονομικές συνέπειες είναι τραγικές, έχουν μολυνθεί ακόμα και τα νεαρά δένδρα και δυστυχώς ε, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό με πιο συνολικό τρόπο λαμβάνοντας υπόψη και τον κατεπήγοντα χαρακτήρα. Λοιπόν, ετούμεθα ένα πρόγραμμα δράσης άμεσο και σε επίπεδο έρευνας, διότι δεν έχουμε λύσεις για να μπορέσουμε να παρέμβουμε αποτελεσματικά. Να υπάρξει σαν παράδειγμα μια επιλογή ορισμένων ειδών ελαιοδένδρων πιο ανθεκτικών στο βακτήριο αυτό για να αποφύγουμε και την διάδοσή του σε άλλες περιοχές. Η Γενική Διεύθυνση Έρευνας λοιπόν θα πρέπει το ταχύτερο δυνατό να βρει μια λύση όπως το έχει κάνει στο παρελθόν σε αντίστοιχες συγκεκριμένες καταστάσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. E, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματος της ομάδας των συντηρητικών, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας επίτροπε. Είστε υπεύθυνο ε, για ένα πολύ σημαντικό τομέα για την ε, λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που άπτεται και της γεωργίας και γενικότερα των τροφίμων και της ασφάλειας των τροφίμων Αναφερθήκατε σε επιμέρους θέματα και αναφερθήκατε επίσης και στον χείριο πυρετό. Θα ήθελα εδώ να μου δώσετε ε, κάποιες διευκρινήσεις. Μας λέγουν ότι η ζωονόσος αυτή προέρχεται από τη Ρωσία. Αλλά το εμπάργο είναι αντίστροφο, δηλαδή απαγορεύεται η εισαγωγή κρεάτων χείρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Ρωσία. Τι περίεργη κατάσταση είναι αυτή. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αντιδράσει ικανοποιητικά. Ε, επίσης τι γίνεται με τις επιδοτήσεις προς τους γεωργούς. Μέχρι τώρα οι προσπάθειες αποζημίωσης των γεωργών ήταν ιδιαίτερα περιορισμένες. Οι ε, κτηνοτρόφοι στην Ανατολική Ευρώπη, κυρίως στην Ανατολική Ευρώπη, έχουν ανάγκη από βοήθεια γιατί μόνοι τους δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Ε, το δεύτερο αφορά τις λεγόμενες ε, τελετουργικές σφαγές. Ε, ξέρετε ότι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν απαγορεύεται η τελετουργική σφαγή ζώων. Θα πρέπει οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν την επιλογή. Κάποιοι θα πρέπει όμως να έχουν την επιλογή και να μην καταναλώνουν ε, προϊόντα κρέατος που προέρχονται από τελετουργικές φαγές. Πρέπει να δοθεί δηλαδή η δυνατότητα επιλογής. Α, και μία τρίτη ερώτηση και αναφέρεται στη στήρωση των χείρων. Ε, εδώ ε, ακούσαμε ότι το 2018 θα πρέπει να τεθεί τέλος στη χημική στήρωση και να υπάρξουν εναλλακτικές λύσεις. Πού έχετε φτάσει, σε τι προτάσεις καταλήγετε. Eh, Ο κύριος Πόλσεν, πρόεδρε, ευχαριστώ. Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω εδώ, κύριε Επίτροπε, για να συζητήσουμε για τα θέματα της μικροβιακής αντίστασης. Είναι ένα θέμα που με ανησυχεί ιδιαίτερος, διότι ασχολούμαι με την έκθεση για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Δεν υπάρχει λόγος να σας εξηγήσω τώρα γιατί είναι τόσο σοβαρό το θέμα αυτό. Το είπατε και εσείς ο ίδιος. Ωστόσο, τώρα που αντιμετωπίζουμε με ενιαίο τρόπο την αλυσίδα παραγωγής, θα ήθελα να σκεφτούμε και τη δυνατότητα μιας πολιτικής ε, μέρημνας για τα ζώα που να είναι και αυτή ενιαία δεν μπορούν όλα να λύνονται, Επίτροπε, με την ε, επικουρικότητα. Για να αποφύγουμε τον αθέμητο ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά, πρέπει να έχουμε αυτή την ενιαία προσέγγιση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να υπάρχει και μια σταθερή θέση στι διαπραγματεύσει μα με του Αμερικανού. Ακόμα και στι ΗΠΑ αυτή τη στιγμή αρχίζει μια εντονότατη συζήτηση ώστε τα ζώα να μην λαμβάνουν ε, αντιβιωτικά κατά την εκτροφή τους και παρόμοια με την, ευρωπαϊκή συζήτηση για την καλύτερη μεταχείριση προς τα ζώα. Οι κτηνοτρόφοι, ό,τι συμφωνίες και αν συνάψουμε με τους Αμερικανούς για τι ελεύθερε συναλλαγές, θα πρέπει να ακολουθούν τα υψηλά μας πρότυπα για την εκτροφή των ζώων. Θα πρέπει να υπάρξουν αυστηροί νόμοι για τη χρήση των αντιβιωτικών που να προβλεφθούν ταυτόχρονα με την παρόμοια νομοθεσία που θα υιοθετήσουν οι Αμερικανοί. Ας μην ξεχνάμε και αυτή την ε, παροιμία ότι ένα χαρούμενο γουρούνι μπορεί να μας δώσει και καλό κρέας και να κάνει τον κτηνοτρόφο του να χαίρεται, το χειροπαραγωγό. Ευχαριστούμε πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβαση η κυρία Σάβανα. Ευχαριστώ, gracias, presidente. Gracias, comisario. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον κύριο Επίτροπο που μας κατέθεσε τις προτεραιότητές του και τις προτάσεις του για τους επόμενους μήνες. Υπάρχουν πολλά πράγματα πάνω στα οποία θα ήθελα να θέσω ερωτήσεις, αλλά θα περιοριστώ υπο, ε, υποχρεωτικά στα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα. Θα ήθελα να μάθω τι μέτρα θα πάρετε για να μην υπάρξει επιμόλυνση των γειτονικών καλλιεργητών. Οι χώρες οι οποίες θα περάσουν από τη διαδικασία αδειοδότησης καλλιέργειας τροποποιημένων γενετικά προϊόντων, τι εγγυήσεις θα δώσετε στις γειτονικέ καλλιέργειες ότι δεν θα μολυνθούν. Υπάρχει επίσης ε, το πρόβλημα με το μέλι. Ε, πώς θα προστατεύσετε τις μέλισσες από τη μόλυνση από γενετικά τροποποιημένα και επίσης πώς θα εμποδίσετε την επιμόλυνση από τη μία χώρα στην άλλη. Είχαμε πει ότι δεν θα υπάρξουν υποχωρήσεις στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων. Συνεπώς θα ήθελα να μάθω στην περίπτωση που υπάρξει έγκριση του TTIP και επιβεβαιωθεί η συμφωνία με τον Καναδά, αν θα υπάρξει μηχανισμός απαγόρευσης εισαγωγής κρεάτων από τη ΣΥΠΑ και τον Καναδά και προϊόντων κρέατος που προέρχονται από ζώα που έχουν καταναλώσει ορμόνες, στα οποία έχουν χορηγηθεί ορμόνες, όπως επίσης και προϊόντα κρέατος που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα. Äh, Ευχαριστώ, Επίτροπε. Ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα εδώ. Μιλήσαμε για την ε, αντιμικροβιακή αντίσταση και στο πακέτο για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Δεν βλέπω καμία ιδιαίτερη διάταξη για τον περιορισμό της χρήσης των αντιβιωτικών. Ε, μας ενδιαφέρει αυτό πάρα πολύ για τη φάση της εκτροφής των ζώων. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει όχι απλώς να μιλήσουμε γενικόλογα, αλλά να έχουμε ελάχιστη χρήση των αντιβιωτικών. Έπειτα για τα φυτοφάρμακα. Μιλήσατε για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Φοβάμαι ότι εν ώψη του TTIP η όλη διαδικασία θα οδηγηθεί σε καθυστέρηση. Είπαμε ότι έπρεπε να βρεθεί μια λύση πριν το τέλος του 2012 αρχικά, αλλά δεν θα έλεγα ότι αυτό που ζήτησε το Κοινοβούλιο έγινε σεβαστό ακριβώς. Από ό,τι ακούστηκε, το γλυφοζάτ έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο των ε, καρκινικών ουσιών, των ε, καρκινογόνων ουσιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό και επίσης τι έχετε να πείτε για τα γάμματα φόμικρων, γιατί στις 22 Απριλίου λέτε υπάρχει μια πρωτοβουλία που προβλέπετε. Μπορείτε να μας δώσετε μια πρόγευση, λίγες λεπτομέρειες γι' αυτό, ε, στα πλαίσια του δημοκρατικού ελέγχου που αποτίθεται ότι θα ασκήσουμε. Ε, όπως τα ξέρετε, τα ε, Εθνικά Κοινοβούλια σας ενημερώνουν για την κατάσταση στην Ευρώπη. Θα σας θυμίσω ότι είναι πολύ τερογενής και τερόκλητη η υλοποίηση και η μεταφορά των ε, οδηγιών αυτών από κράτος σε κράτος. Σας, σας ευχαριστώ που ήρθατε να μιλήσετε και για τους, ε, και για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες είναι ένα πρόβλημα και είναι ένα πρόβλημα ήδη από πολύ παλιά όταν άρχισα να ασχολούμαι από το 1967. Εγώ είχα χρησιμοποιήσει τότε ουσίες και δεν είχα προστατευθεί αλλά εξακολουθώ να υπάρχω σήμερα. Αν απαγορευθούν αυτοί, αυτές οι ουσίες φοβάμαι ότι πάρα πολλά όπλα που έχει κανείς εφόσον είναι αγρότης για να καταπολεμήσει τα αγριόχωτα κτλ θα εξαφανιστούν και ε, θα έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα. Αλλά αν πράγματι λοιπόν απαγορευθούν στη φυτική παραγωγή θα έχουμε πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα και δεν θα έχουμε καλλιέργειες και θα εισάγουμε τα προϊόντα από τρίτες χώρες που τα χρησιμοποιούν. Θα ήθελα να υπενθυμίσω την Επιτροπή μας ότι η Υπηρεσία Ασφάλειας της Φυτικής Παραγωγής δεν θεωρεί ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στον τομέα αυτό. Η έκθεση στα εντομοκτώνα γενικά και σε αυτά τα προϊόντα είναι ένα πρόβλημα, αλλά όχι όμως ιδιαίτερα υψηλό. Τώρα για το καμπυλοβακτήριο. Ε, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελεγχθεί το θέμα ε, του ε, καμπυλοβακτηρίου στην παραγωγή, στην ορνηθοπαραγωγή. Πρέπει να υπάρξουν κάποιες ρυθμίσεις, αλλά σε χώρες όπως η Δανία που τα πάνε αρκετά καλύτερα θα το αντιμετωπίσουν, ενώ οι μεσογειακές χώρες θα έχουν πάρα πολύ σοβαρά θέματα να αντιμετωπίσουν. Η λύση βρίσκεται όμως σε αυτόν ο οποίος μαγειρεύει το κοτόπουλο. Αν το μαγειρεύει σωστά, κανένα πρόβλημα με το καπυλοβακτήριο. Με ευχαριστώ πολύ. Ένα λεπτό τώρα πλέον οι συνάδελφοι. Η κυρία Χέρενς Γαρσία. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για την παρουσία του και θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση σχετικά με τη ζώνος. Έχουμε την ξυλέλια φαστιζιώσα, έχουμε επίσης και άλλα προβλήματα τα οποία επηρεάζουν τη φυτική παραγωγή διορθώνω. Ε, μπορεί να υπάρξει ένας θετικός κατάλογος χωρών και περιοχών που, αντιμετωπίζουν, που δεν αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα έτσι ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε ε, σχέσεις ε, ανταλλαγής εμπορικών στοιχείων, εμπειριών κτλ. Υπάρχει μια κάποια τεχνολογία ε, η οποία να είναι ικανοποιητική. Είμαστε υποχρεωμένοι να προσφύγουμε στα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα. Θέλουμε πιο συγκεκριμένες προτάσεις, ε, επίσης ε, και για τους τρόπους ελέγχου θα υπάρξει μια εθνικοποίηση με διαφορετικά επίπεδα προστασίας και ελέγχου. Πιστεύετε ότι θα ήταν ιδιαίτερος επικίνδυνο για την ενιαία αγορά και κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε ιδιαίτερες εμπορικές τρευλώσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαπραγματεύσεις με την Ιαπωνία. Αρμοδιότητας δική σας. Υπάρχει περίπτωση η Ιαπωνία να σεβαστεί την περιφερειοποίηση που έχουμε υιοθετήσει. Γιατί υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν μπορούν να εξαγάγουν στην Ιαπωνία σήμερα λόγω του ε, προβλήματος της πανόλης των χείρων. Ο κύριος Μπιόρκ μας είπε ότι ήθελε η Επιτροπή να επανεξετάσει το σύνολο μέτρων για την ε, υγιεινή και μας έλεγε ότι πρέπει για τη και μας έλεγε ότι πρέπει να υπάρχει ε, υπάρχουν όροι για την σφαγή στα, στις μονάδες εκτροφής τέτοιοι που να περιορίζουν τον αριθμό των ενδιαμέσων στην αλυσίδα της σφαγής. Ε, έχετε σε αυτό κάτι να πείτε. Μια άλλη ερώτηση. Έχουμε κοινέ φυτοϊγειονομικές διατάξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δηλώσεις. Αυτό πόσο έχει προχωρήσει προς το παρόν. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ, κύριος Χάζελκαγκ. Eh, Κυρία Χάζελκαγκ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που ήρθατε. Έχετε όντως μια σειρά από σχετικά ζητήματα, την μικροβιακή αντοχή, απόβλητα κουζίνας, τροφίμων, ε, μάλλον ε, αποτελέσματα της συμπεριφοράς και του τρόπου του εντατικού της εκτροφής που έχουμε υιοθετήσει. Η εντατικοποίηση όμως βλέπουμε δυστυχώς ότι συνεχίζεται. Και βλέπουμε ότι τα ζώα συνοστίζονται ε, και μεταφέρονται μαζικά από την μια άκρη στην άλλη της Ευρώπης. Διαρωτώ με λοιπόν, η δική σας θέση σε σχέση με την εντατικοποίηση του γεωργικού τομέα στην Ευρώπη ποια είναι. Στις κάτω χώρες βλέπουμε παραδείγμα ότι, ότι αναπτύσσονται επιζωοτίες στις κάτω χώρες βλέπουμε ότι οι ακριβώς αναπτύσσονται στις περιοχές εντατικοποίησης γεωργικής εκτροφής. Συμφωνείτε ότι οι ε, επιδοτήσεις της γεωργίας πρέπει να καταργηθούν. Ο Πρόεδρος. Καπούτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ Επίτροπε, όχι μόνο για την παρουσία σας εδώ, αλλά για την στάση την οποία φαίνεται ότι διαμορφώνεται απέναντι ε, στον διάλογο που πρέπει να υπάρχει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μετά από τις συζητήσεις που έχουν γίνει στην ε, Ολομέλεια ε, για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Θα δούμε με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα στο μέλλον. Και εγώ όμως θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με την αντίσταση στα αντιβιωτικά να προσθέσω μάλλον κάποια στοιχεία σε αυτά τα οποία είπε η συνάδελφος Πάουλσεν και τα οποία είναι πράγματι εξαιρετικά. Θα ήθελα να καταλάβω τι σκέφτεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι επιπτώσεις οι αρνητικές των αντιβιωτικών είναι πλέον σαφείς. Υπάρχουν κάποια προγράμματα από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να υπάρξει σωστή και υπεύθυνα προσανατολισμένη χρήση τουλάχιστον των μορφών αντιβιωτικών που χρησιμοποιούνται κυρίως και στην ιατρική για τον άνθρωπο αλλά και στην κτηνιατρική θα ήθελα να αποφύγουμε οι κτηνίατροι να πολλούν οι ίδιοι τα φάρμακα, γιατί αυτό συμβαίνει σε ορισμένες χώρες. Έχουμε βέβαια την εξαίρεση της Δανίας, στην οποία έχει υπάρξει μια σημαντική μείωση της πώλησης και κατανάλωσης αυτών των φαυσιών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος ομιλητής Αφού σας ζητήσω όμως ε, να είστε σύντομοι. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, μια ερώτηση για την κλωνοποίηση, λέει η κυρία Μύρα. Και για το θέμα της ε, επισήμανσης τροφίμων σε περίπτωση χρήσης ε, κλωνοποιημένων προϊόντων, των εισαγωγών τους και βέβαια τις διαπραγματεύσεις της TTIP. Και έχω επίσης θέματα για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Και για είδη επεκτατικά όπως ο δάκος του κερασιού και αντίστοιχα ε, τέτοια ε, παράσιτα θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω ποια είναι η κατάσταση, αν την παρακολουθείτε και τι έχετε διαπιστώσει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Έχω και εγώ μια σειρά από ερωτήσει. Έχουμε χρησιμοποιήσει πολλά ζώα, πολλά είδη, λέει ο κύριο Γιάρ, για τα αντινικοτιοειδή παραδείγματι, υπάρχουν κάποιε αξιολογήσει και θέλουμε να δούμε αν έχετε καταλήξει κάπου σε σχέση με τις συνέπειες τη δημόσια υγεία και τη γεωργία ασφαλώς και αν οι γεωργοί ενημερώνουν ε, ποια προϊόντα μπορεί να χρησιμοποιήσουν στις επόμενες περιόδους για τα αντιβιωτικά. Υπάρχουν ε, αντιβιωτικά τα οποία μπορεί να χρησιμοποιούνται μόνο στον άνθρωπο ή και στη γεωργία. Έχετε κάποια εικόνα συγκεκριμένη για το ποια είδη είναι αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Η ε, κυρία Χόιμπουχ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε για την ε, προστασία των ζώων και τη σχετική μονάδα της Γενικής Διεύθυνσης για την Υγεία. Ε, αληθεύει ότι έχει διαλυθεί η σχετική μονάδα και ότι έχουν υπαχθεί αρμοδιότητες σε άλλες, δηλαδή δεν υπάρχει ειδική μονάδα που να ασχολείται με την προστασία της υγείας των ζώων και επίσης για την ε, γενετική μηχανική υπάρχει νέα μελέτη η οποία αξιολογεί τις ε, μελέτες της ΕΦΣΑ για τις ε, μέλισσες που αποδεικνύεται ότι ταξιδεύουν όχι μόνο μερικά μέτρα αλλά χιλιόμετρα. Ερωτώ λοιπόν συγγνώμη, για τις, ε, ναι, για τις οι οποίες μπορούν να μεταφέρουν την γύρι από το γενετικά τροποποιημένο καλαμπόκι για χιλιόμετρα. Ε, θέλω να ρωτήσω αν έχουν αξιολογηθεί οι σχετικοί κίνδυνοι και αν υπάρχει πρόθεση για εισαγωγή νέων ε, διατάξεων από την ΕΦΣΑ, στο πλαίσιο της ΕΦΣΑ καλύτερα, σχετικά με την ε, κυκλοφορία αυτών των ειδών. Ευχαριστώ πολύ. Eh, Κύριος Μπόγκοβιτς, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, εφέτος μία από τις κύριες δραστηριότητες που θα σας απασχολήσουν είναι και οι δραστηριότητες σχετικές με τη διαπραγμάτευση της TTIP, της Διατλαντικής Εμπορικής Συμφωνίας και Συμφωνίας για τις Επενδύσεις. Ε, σε αυτό θα εστιαστώ εγώ. Έχουν ακουστεί πολλές επικρίσεις για την απουσία διαφάνειας στις διαπραγματεύσεις αυτές. Διάφορα έγγραφα ε, φαίνεται να ανταλλάσσουν χέρια και κλεισμένων των θυρών ή μπορεί κανείς να τα διαβουλευτεί ως βουλευτής, να τα συμβουλευτεί ως βουλευτής μέσα σε κλειστά δωμάτια. Εγώ έχω καταφέρει να μελετήσω κάποια αυτά έγγραφα, αλλά διαιρωτώ με, όταν τεθεί σε εφαρμογή τη TIP στην Ευρώπη, θα εξακολουθεί να απαγορεύεται η χρήση η εισαγωγή στην Ευρώπη κρέατος ε, με ορμόνες. Για τα ζυζανιοκτώνα υπάρχει περίπτωση να ε, προκύψουν αλλαγές ως προς την ε, νομοθεσία και τι είδου ζυζανιοκτώνα θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε στην Ευρώπη, θα διαφυλαχθούν δηλαδή οι ψηλές προδιαγραφές που έχει ορίσει στο παρελθόν η Ευρώπη. Αυτά όλα τα ρωτάω, διότι με ενισχύει ιδιαίτερα το γεγονός ότι εάν δεν μπορέσουμε να επιδείξουμε στάση σοβαρή και υπεύθυνη για να δώσουμε απαντήσεις εγκαίρως στα προβλήματα αυτά, η TTIP μπορεί να αποτύχει λόγω αυτών ακριβώς των συστημάτων και πρέπει να καθησυχάσουμε τον καταναλωτή, τον Ευρωπαίο καταναλωτή, ότι δεν θα υποβαθμιστούν τα πρότυπά μας. Ευχαριστώ κυρία... ο κύριος Λουαζού. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ασφάλεια στο τρόφιμα θα υπάρξει αν δεν, είμα, έχουμε και την ελευθερία και την κυριαρχία συνώνυμες αυτής της ε, ασφάλειας των τροφίμων. Είδαμε τις ε, υπερβολικά, τις άκρατα φιλελεύθερες πολιτικές που επιδιώκουν το κέρδος εις βάρος της ποιότητας τα τελευταία χρόνια να μας φέρουν στην κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε τώρα με όλους τους κινδύνους ε, ενώ ζητάμε ε, επισήμανση, επισήμανση πάνω απ' όλα γιατί τη διεκδικεί ο καταναλωτής που έχει βαρεθεί πια να τρώει ό,τι να είναι. Ε, η εκδήλωση διατροφικού πατριωτισμού και επιλογής τοπικών προϊόντων θα έπρεπε να αποτελέσει ένα μήνυμα αφύπνισης Πρέπει λοιπόν να προχωρήσετε με ε, αποφάσεις οι οποίες δεν θα εξωτερώνουν την ε, εθνική κυριαρχία, δεν θα επιδιώκουν μόνο το οικονομικό κέρδος και θα εξασφαλίσουν διατροφική ασφάλεια. Δεν έχει έρθει πια η ώρα να αλλάξετε πολιτική. Ο κύριος Ταραμπελά. Μεταξύ όλων των τόσο ενδιαφερόντων θεμάτων που θίξατε κύριε Επίτροπε, ήταν όλα πολύ σημαντικά, Δύο θέλω να θίξω. Ένα, την επενσήμανση των ε, προϊόντων κρεατός, για τον οποίο καταφέραμε μεγάλη πρόοδο, όμως για τα ήδη προετοιμασμένα γεύματα δεν έχουμε ε, κάνει μεγάλη πρόοδο. Μιλήσατε για την μελέτη που παρουσιάστηκε από τις εταιρείε παραγωγής τροφίμων. Οι καταναλωτές έχουν την ε, δική τους άποψη. Είδαμε την εμπειρία της Γαλλίας με το επιπλέον χρέος, ε, κόστος να είναι στο 0,02%. Δεν είναι και πολύ σημαντικό και συζητήσαμε και στο Στρασβούργο τα θέματα αυτά Βαίνεται ότι υπάρχουν αντιστάσει που βασίζονται στα επιχειρήματα των εταιριών και αυτό είναι όλο. Οπότε α είμαστε λίγο πιο προπαντιστέ και να προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε για του καταναλωτέ παγκοσμίω. Έπειτα για την κλεινοποίηση και εδώ το συζητήσαμε αρκετά πρόσφατα και φάνηκε ξεκάθαρα ότι είναι ακριβό, υπάρχουν κίνδυνοι, προβλήματα για την υγεία και την ευζοία των ζώων Κανείς δεν την θέλει. Γιατί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, το κλείνει το θέμα αυτό, να το βάλει στο χρονοτούλαπο και να πει δεν θέλουμε την κλωνοποίηση, να είναι ξεκάθαρο. Στα, μέρη, στα πλαίσια της καλύτερης νομοθεσίας θα είναι η καλύτερη νομοθεσία, η βέλτιστη που θα μπορούσατε να προβλέψετε. Ευχαριστώ. Η κυρία Νόχλ, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε. Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει ένα νέο χρονοδιάγραμμα και νέα πρόταση για το γενετικό υλικό στο τραπέζι σας και αν έχετε κάτι να μας ανακοινώσετε. Θέλω να σας υποστηρίξω στο, στη σαφή τοποθέτηση για τα πρότυπα στον χώρο των τροφίμων. Ότι δηλαδή δεν πρόκειται να υπάρξουν ε, υποχωρήσεις στην TTIP ως προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Είπατε τη λέξη υποχωρήσεις και χαίρομαι ιδιαίτερως γι' αυτό. Ότι θα ακολουθήσετε μια σκληρή και σαφή γραμμή. Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να σταθούμε ενωμένοι για να διαφυλάξουμε τις προδιαγραφές μας και τον τρόπο ζωής μας. Ευχαριστώ πολύ, Άντριου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε σειρά μου να θέξω από τα σημαντικά ζητήματα που τέθηκαν. Δύο που θέλω να, σε δύο θέλω να σταθώ. Ήχνη λασιμότητα και πρέπει να το πούμε με πολύ ε, ένταση ότι για τα παρασκευασμένα γεύματα, τουλάχιστον το 97% των καταναλωτών το ζητούν, εμείς το ζητούμε, οπότε εξηγήστε μας γιατί έχετε ε, επιφυλάξεις για την επισήμανση στο κρέας και στα προπαρασκευασμένα γεύματα. Ξέρετε ότι ήδη από το 2013 έχουν αμφισβητηθεί οι προτάσει σα. Δεν πρέπει να δούμε ε, την εμπιστοσύνη των καταναλωτών ω βασικό μέρο του προβλήματο. Και έπειτα το θέμα των, ε, του βακτηριδίου που πλήττει τα ελαιόδεντρα. Ξέρετε τι γίνεται με τον έλεγχο των ε, φυτών που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από όσε ανησυχίε υπάρχουν εκεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μέχρι τώρα ήταν κατηγορηματικά αντίθετη. Μήπω πρέπει να αλλάξει τη διαδικασία των ελέγχων που για τι εισαγωγέ προ την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί η κλεψιέλα προστίθεται σε άλλα παράσιτα όπως τον δάκο των λιόμαντρων και προβλέπονται ε, τεράστιες ζημιές στον τομέα της ολοπαραγωγής. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για τις διευκρινήσεις που έδωσα για, το, για τις εισαγωγές χείριου κρέατος προς τη Ρωσία. Ξέρουμε ότι το 50% του ΑΕΠ μας έχει μειωθεί λόγω της χρήσης των αντιβιωτικών. Όμως, εκτινοτρόφοι ε, και όλοι οι ενδιαφερόμενοι θεωρούν ότι πρέπει να μειωθούν ε, κι άλλο τα αντιβιωτικά στη χρήση για να μην υπάρξει περαιτέρω υποβάθμιση της υγείας των ζώων. Ήθελα λοιπόν τη δική σας γνώμη. Ο υφυπουργό μας ε, ζήτησε να διεξαχθούν σχετικέ μελέτες Οπότε είναι σαφές ότι πρώτη προτεραιότητα πρέπει να είναι η δημόσια υγεία. Όμως υπάρχει ένα δίλημα. Τι θα κάνουμε. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι και να μειώνουμε τη χρήση των αντιβιωτικών ε, εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις ε, νόσους. Τις Δεν μπορούμε να πλήξουμε την ανθρώπινη υγεία εδώ. Πού βρίσκεται το σημείο ισορροπίας. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ τον Επίτροπο που ήρθε και για τις πολύ διεξοδικές του εξηγήσεις. Έχω μια, δύο ερωτήσεις, καταρχάς για τα αντιβιωτικά που χρησιμοποιούνται στην κοινοτροφία. Το ανέφερε και ο κύριος Δέσνο νωρίτερα ότι η Γερμανία έχει ένα πολύ, περίπλοκο, ένα πολύ πλήρες και περίπλοκο σύστημα παρακολούθησης. Είναι γνωστό δηλαδή πού, σε ποιο σημείο, πότε και ποιο ζώο έχει λάβει αντιβιωτικά ως θεραπεία. Εδώ λοιπόν με την TTIP Θα πρέπει μάλλον να προβλέψουμε ένα πανευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης για να είμαστε σε θέση να αντιδρούμε αμέσως. Το άλλο ζήτημα έχει να κάνει με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Ε, ήσασταν άλλωστε παρόν και εσείς στις διαπραγματεύσεις και θέλω να σας ευχαριστήσω ρητά γι' αυτό. Μπορούμε να έχουμε δηλαδή μια καλή ε, ρύθμιση για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, αλλά παραμένει το ζήτημα της ε, της οικολογικής ε, γεωργίας και της ε, παρουσίας γενετικά τροποποιημένων οργανισμών όπου θα ήθελα να ρωτήσω τι είδους επισήμανση μπορούμε να προβλέψουμε εκεί. Τι έχει να πει η Επιτροπή σε αυτό. Ευχαριστώ, Σεμπαστιά. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Κάποιες ερωτήσεις σχετικές με την ευημερία των ζώων. Όλα τα κράτη-μέλη δεν έχουν εφαρμόσει πλήρως την, τον αρμόδιο κανονισμό, εν πάση περιπτώσει, τον σχετικό με την ευημερία των, των ζώων. Υπάρχουν πολλά προβλήματα και σε σχέση ε, με τα πουλερικά και σε σχέση με άλλα ζώα υπάρχουν προβλήματα και για τη θανάτωση και στο επίπεδο της θανάτωσης όπως επίσης και στο επίπεδο της μεταφοράς τους. Έχετε ξεκινήσει την πρωτοβουλία για τον περιορισμό της μεταφοράς σε 8 ώρες πριν υπάρξει μια διακοπή. Έχουμε προβλήματα στην Ισπανία και με την παραγωγή τώρα ελαιολάδου όπως επίσης και με την παραγωγή εσπεριδοειδών και υπάρχει η γνωστή, μια γνωστή ασθένεια η οποία έχει έρθει από τη Βόρεια Αφρική. Τι μέτρα σκοπεύετε να πάρετε για αυτή την ασθένεια από την Βόρεια Αφρική. Ε, Ο κύριος Δόρμαν. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την TTIP. Ήμουν στην Ουάσιγκτον με την αντιπροσωπεία μας εκεί, στο Κογκρέσο, όπου διαπίστωσα ότι δεν είναι διατεθειμένοι οι Ευρωπαίοι, να, οι Αμερικανοί να δουν την Ευρώπη ως μια ένωση και ότι προσπαθούν να ε, ξεχωρίσουν τα κράτη-μέλη και να διαπραγματεύονται με το κάθε ένα χωριστά. Φερρυπίν, για το βόηο κρέας ε, εξαγωγές δέχονται μόνο από την Ιρλανδία, για τα μήλα και τα χλάδια από 8 κράτη-μέλη συγκεκριμένα και όχι από άλλα. Και βλέπουμε ότι σε σχέση με την ασφάλεια των ε, τροφίμων, τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε εμεί στην Ευρώπη θα είναι σημαντικότερα από αυτά που θα έχουν να αντιμετωπίσουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Εμεί τώρα εισάγουμε μήλα από το Wisconsin και την Καλιφόρνια και όχι από άλλες ε, πολιτείες. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω αν σας έχει απασχολήσει το θέμα αυτό και αν έχετε αναζητήσει λύσεις ε, και διεξόδους για τις εξαγωγές μας. Παράλληλα όμως μαζί με το θέμα της ασφάλειας των τροφίμων. Σας ευχαριστώ. Domnule comisar, ați vorbit foarte bine despre pesta porcină, Ευχαριστώ Πρόεδρε, μιλήσατε για το χείριο κρέας, μιλήσατε για νόσο των πουλερικών, αλλά και για το βακτηρίδιο που πλήττει τα ελέγχοντρα. Έχετε κάποια ε, στρατηγική για τον αυθόδη για την όσο των ε, βοηδών ε, θα πρέπει να το δούμε για Επίσης και γιατί αυτό μας ε, διαταράσσει και τις συναλλαγές με τη Ρωσία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον ε, ε, κύριο Επίτροπο που είπε πολλά θετικά πράγματα. Με ενδιαφέρον τα άκουσα. Εγώ είμαι ε, αρμόδια, είμαι εισηγήτρια για τα θέματα των φυτοφαρμάκων και με ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτά τα οποία είπε. Παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια τροποποίηση του κανονισμού 226 ε, του 2004 σχετικά με την αδειοδότηση και τον έλεγχο των κτηνιατρικών προϊόντων που, των οποίων ο έλεγχος θα πρέπει να φτάσει στο ίδιο επίπεδο με τα, τον αντίστοιχο τρόπο αδειοδότησης των φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπους. Έτσι θα διασφαλίσουμε και θα αυξήσουμε την ποιότητα των κτηνιατρικών φαρμάκων γιατί τελικά προκαλούν, μπορεί να προκαλέσουν τα ίδια προβλήματα που προκαλούν και τα φάρμακα στον άνθρωπο. Και τι γίνεται ακριβώς με την υπηρεσία που θα ασχοληθεί με τα ακτινιατρικά φάρμακα, τι εξηγήσει μπορείτε να δώσετε για την αδράνεια τη οποία έχει σημειωθεί. Γιατί δεν ε, έχετε προχωρήσει νομοθετικά. Δεν έχουμε καταλάβει ακόμα Τελειώνοντας τώρα, μια και είμαι Ισπανίδα, έχουμε το πρόβλημα με τα ελαιόδένδρα. Τα είπαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι. Ε, τι ε, προσκοπεύετε να κάνετε στο μέλλον για την ασθένεια αυτή των ελαιοδένδρων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο, λέει ο κύριος Φέντερ λέει, γιατί αναφέρθηκε σε ένα πολύ σοβαρό θέμα όπως είναι η αντίσταση στα αντιβιωτικά. Συζητήσαμε πολλά θέματα σήμερα εδώ, παρόλα αυτά ίσως να πρέπει να διαβρύνουμε ακόμα περισσότερο το πεδίο μας. Ε, τι πρέπει να κάνετε σε διεθνές επίπεδο, σε επίπεδο συνεργασιών. Υπάρχουν πάρα πολλοί και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φορείς ενώ, που θέλουν να μετριάσουν την κατανάλωση των αντιβιωτικών. Αλλά ξέρουμε ότι μια πραγματικά άκρατη χρήση των αντιβιωτικών δεν συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά σε χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία. Μπορείτε λοιπόν να κάνετε κάτι έτσι ώστε να επηρεάσετε τα πράγματα και σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεύτερο ερώτημα, θα ξεκινήσετε πρωτοβουλίες ή ξεκινάνε μάλλον πρωτοβουλίες για την δημιουργία νέων τύπων προχωρημένων αντιβιωτικών. Ε, πώς θα μπορέσετε ε, να ελέγξετε την κυκλοφορία τους καλύτερα. Σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Ακούσαμε πράγματι όλους όσους ήθελαν να θέσουν ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ όλους για τη συνεισφορά σας και τη συντομία σας. Δεν ευχαρίστησα τον καθένα ξεχωριστά για να κερδίσουμε χρόνο δίδω το λόγο στον Επίτροπο Αντροκάτης. Α, υπάρχει ένα θέμα επιπλέον το οποίο αφορά την ξυλέλεια, ε, το γνωστό βακτήριο για τα ελαιόδενδρα. Θα τεθεί το θέμα αυτό αργότερα. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα δεν μπορώ να δώσω απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικές οι ερωτήσεις αυτές και απαιτούν οι περισσότερες λεπτομερείς απαντήσεις. Για το θέμα του βακτηρίου που έχει χτυπήσει την ελαιοπαραγωγή, άλλωστε θα ακολουθήσει μετά από μένα μια συζήτηση εδώ με ειδικού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα περάσουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες για το βακτήριο ξυλέλια. Θα ήθελα για τις περισσότερες ερωτήσεις οι οποίες έχουν τεθεί να απαντήσω και γραπτός έτσι ώστε ε, να λάβω υπόψη μου πολύ περισσότερα συγκρετημένα στοιχεία και να δώσω τεκμηριωμένες απαντήσεις. Αλλά θα δώσω κάποιες απαντήσεις τώρα εδώ, ξεκινώντας με τις πρώτες ερωτήσεις. Η ερώτηση του κυρίου Ντες. Αναφερθήκατε στην αντιμικροβιακή αντίσταση, στην, αντιβιωτική, στην αντίσταση στα αντιβιωτικά. Εγώ είμαι γιατρός και δεν μπορώ παρά να υπογραμμίσω το τεράστιο πρόβλημα που δημιουργεί η αντίσταση στη χρήση των αντιβιωτικών. Εγώ θα ήθελα και ε, το θέμα να το δούμε από δύο πλευρές και από πλευράς της ανθρώπινης κατανάλωσης άμεσα αλλά και από πλευράς της χρήσης των αντιβιωτικών σε κτηνιατρικό επίπεδο. Νομίζω ότι απαιτείται μια στρατηγική αντίληψη για την χρήση των αντιβιωτικών. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το σύνολο της αλυσίδας από τα ζώα μέχρι τους ανθρώπους. Ε, βασική ιδέα είναι να προσπαθήσουμε να καταγράψουμε με σωστό τρόπο, με κοινό τρόπο όλες τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε και για την κατανάλωση απευθείας από ανθρώπους και για την κατανάλωση έμεσα από τα ζώα. Προσπαθούμε να αναθεωρήσουμε το πρόγραμμα δράσης μας, το οποίο έχουμε εδώ και μία πενταετία. Ξέρετε ότι στις 26 Φεβρουαρίου του 2015 κυκλοφόρησε μια έκθεση η οποία παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας που έχει γίνει μέχρι τώρα. Θα θέλαμε λοιπόν να αναπτύξουμε μια συνολική στάση απέναντι στην χρήση ε, των αντιβιωτικών σε όλα τα επίπεδα. Ε, προφανώς θα ήταν ε, σωστό σε αιτήσια βάση να γίνεται μια καταγραφή και μια δήλωση για την κατάσταση της υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μπορέσουμε δηλαδή να καταλήξουμε σε συγκεκριμένους δείκτες, σε συγκεκριμένα θέματα γύρω από τα αντιβιωτικά, γύρω από τις χρόνιες ασθένειες και να αποκτήσουμε μια κοινή εικόνα, εν πάση περιπτώσει, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έτσι μόνο θα μπορέσουμε να κάνουμε προτάσεις για την ουσιαστική μείωση της χρήσης των αντιβιωτικών. Για να μειωθεί η ποσότητα των αντιβιωτικών δεν χρειάζεται μια απλή παρακολούθηση των, των νοσούντων, αλλά απαιτείται να αλλάξουν και οι μεθοδολογίες αντιμετώπισης των παθολογιών και το ίδιο ισχύει και για τα ζώα. Θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνουμε νέα είδη φαρμάκων, όχι αποκλειστικά αντιβιωτικών ουσιών. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την καινοτομία στις φαρμακευτικές ουσίες Καλό θα ήταν λοιπόν να υπάρξει μια κοινή δράση και εγώ ε, θα συζητήσω το θέμα και στη Γενική Διεύθυνση Υγείας ε, με ε, τους αντιπροσώπους του κτηνιατρικού κλάδου και του ιατρικού κλάδου για να καταλήξουμε σε ένα κοινό πρόγραμμα δράσης. Αναφερθήκατε για κάποια καλά, σε κάποια καλά παραδείγματα στη Γερμανία, στην Ολλανδία. Ε, είδα ποιες είναι οι εξαιρετικά ορθές Ολλανδικές πρακτικές για την καταγραφή των δεδομένων για την κατανάλωση των αντιβιωτικών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Έχουν πολύ αναλυτικά στοιχεία και έχουν επίσης και πολύ αναλυτικά στοιχεία ε, για την παρουσία των αντιβιωτικών ουσιών ε, στα νοσοκομεία. Έτσι μπορούν να καταλήγουν σε σωστές προτάσεις. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε πολύ δραστήριοι στη συλλογή στοιχείων έτσι ώστε να βρούμε πρακτικές λύσεις. Και έτσι θα μειώσουμε τη χρήση των αντιβιωτικών. Τέθηκαν και άλλες πολλές ερωτήσεις από τον κύριο Βοησεχόφσκι για τους τρόπους σφαγής, για τα σφαγεία. Υπήρξε μία έρευνα γύρω από τις λεγόμενες τελετουργικές μορφές σφαγής προφανώς και πρέπει να σεβαστούμε την θρησκευτική ελευθερία, αλλά τα κράτη-μέλη εξακολουθούν να παραμένουν υπεύθυνα στις χορήγησεις αποκλήσεων από τα κτηνιατρικά στάνταρτ τα οποία επικρατούν και είναι καθιερωμένα σε όλες τις χώρες. Έχουμε συλλέξει στοιχεία και έχουμε ακολουθήσει μια στρατηγική επί τη βάση των στοιχείων αυτών και κάνουμε μία μελέτη για την σωστή ενημέρωση του καταναλωτή γύρω από τον τρόπο σφαγής ε, του ζώου. Έχει ολοκληρωθεί ε, πρόσφατα η μελέτη συγκεκριμένη. Στην παρούσα φάση δεν έχουμε ακόμα καταλήξει ε, στο εύρος της χρήσης των τελετουργικών μορφών σφαγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας δυστυχώς είναι ελλειπή και περιορισμένα. Κάποια άλλα θέματα τώρα. σε θέματα υγείας, και υγιεινής στη φυτική παραγωγή έθεσε κάποια ερωτήματα η κυρία Έραντς Γαρσία. Το πρόβλημα της ξυλέλια και πώς μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες καλλιέργειες. Εμείς θα κάνουμε κάποιες προτάσεις προστασίας από την ασθένεια αυτή. Θα προσπαθήσουμε να λειτουργήσουμε προληπτικά ε, και να μειώσουμε έτσι τους κινδύνους. Τα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή προσπαθούν να βρουν κάποιες λύσεις, όπως επίσης ε, και ε, ε, ελέγχουμε τους τρόπους για καλύτερη διαδικασία εισαγωγών προϊόντων φυτικής παραγωγής από τρίτες χώρες. Πρέπει όμως βασικά να εφαρμόσουμε την αρχή της πρόληψης Ξέρω ότι κάποιες χώρες ε, θέλουν ε, ένα κλειστό σύστημα, αν θέλετε, προστασίας της ε, φυτικής τους παραγωγής. Εμείς σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή είμαστε φυσικά υπέρ ενός ανοιχτού συστήματος και θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια συμβιβαστική λύση η οποία μας επιτρέπει να λειτουργούμε με προληπτικό τρόπο όταν αναπτύσσονται κίνδυνοι σε συγκεκριμένες χώρες από τις οποίες εισάγουμε προϊόντα και φυσικά καθ' όλη τη διάρκεια της παρουσίας των κινδύνων αυτών να απαγορεύουμε την εισαγωγή προϊόντων από τις συγκεκριμένες χώρες. Για την κλωνοποίηση τώρα. Να πω ότι η επισήμανση ε, θα πρέπει να είναι σωστή για προϊόντα κρέατος αποκλωνοποιημένα. Το θέμα είναι βέβαια να προστατεύσουμε τα ευρωπαϊκά συμφέροντα σεβόμενοι και το διεθνές νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο καλούμεθα να κινηθούμε. Οι προτάσεις ε, του 2013 από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν έγιναν πλήρως δεκτές. Θα πρέπει να δούμε με πιο πρακτικότερο τρόπο τέτοιου είδους μέτρα ε, θα γίνουν δεκτά. Η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας έχει ξεκινήσει ε, μια μελέτη των ζώων κλωνοποιημένων ζώων και απογόνων κλωνοποιημένων ζώων Και να δούμε σε ποιο βαθμό δημιουργούνται προβλήματα για τις παραδοσιακές κτηνοτροφικές δραστηριότητες από τέτοιου είδου θέματα. Ο κύριος Ταραμπέλα έθεσε το θέμα της ονομασίας προέλευσης. Η ονομασία προέλευσης είναι ένα πολλαπλού, ε, πολλαπλών προβλημάτων θέμα το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ την, τα οικονομικά της ιατρικής παραγωγής. Είναι καθήκον λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διασφαλίσει αποφάσεις οι οποίες να είναι τεκμηριωμένες γύρω από τα θέματα αυτά της σήμανσης των συγκεκριμένων προϊόντων. Ιδιαίτερα στον τομέα της πώλησης ε, προϊόντων ε, προερχόμενων από κρέατα. Δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε επιβαρύνσεις για τους παραγωγούς ε, και επιπλέον κόστος. Είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε δηλαδή την έρευνα ε, για τα θέματα της σήμανσης των προϊόντων κρέατος, αλλά παρόλα αυτά να προσπαθήσουμε να κάνουμε βήματα προόδου σύντομα. Ένα άλλο θέμα που έθεσε η κυρία Πάουλσεν για την αντίσταση στα αντιβιωτικά πάλι. θα πρέπει επίσης να μπορούμε να παρέμβουμε στον τομέα αυτό όπως μπορούμε να παρέμβουμε στην καταπολέμηση των μολυσματικών ασθενειών. Αυτό επηρεάζει φυσικά και την παραγωγή κρέατος, τις κτηνοτροφικές δραστηριότητες και την έλογη χορήγηση τέτοιου είδους αντιβιωτικών ουσιών. Ε, έχουμε την δυνατότητα παρέμβασης, έχουμε μια νέα πρόταση τώρα σχετικά με, ε, ε, με τον έλεγχο και την εποπτεία της χορήγησης αντιβιωτικών προϊόντων και αυτά θα πρέπει να παραμείνουν φυσικά στο εσωτερικό του πλαισίου του κανονισμού για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Είπατε επίσης ε, ότι πρέπει να θέσουμε και το θέμα της αντίστασης στα αντιβιωτικά και σε διεθνές επίπεδο. Μα δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της αντίστασης ε, στα μικρόβια αν ε, δεν θέσουμε το θέμα σε επίπεδο ΠΟΕ. ΠΟΗ, συγγνώμη. όπως επίσης και ε, σε διεθνείς οργανώσεις και διεθνή φόρα για την υγεία των ζώων. Μιλάμε για μεγάλες χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία, η Αργεντινή, η Βραζιλία και η ΙΠΑ. Τίθενται λοιπόν πολλά προβλήματα τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν στα πλαίσια των σχέσεων που έχουμε με τις συγκεκριμένες αυτές χώρες. Έτσι θα ανυψώσουμε ακόμα περισσότερο τα επίπεδα προστασίας των τροφίμων μας. Και σε επίπεδο λοιπόν του Παγκόσμιου ε, Οργανισμού Υγείας μπορούμε να συζητήσουμε το θέμα ιδιαίτερα της αντίστασης στα αντιβιωτικά. Έχουν τώρα πλέον ξεκινήσει οι συζητήσεις τις οποίες παρακολουθούμε γιατί όπως είπατε έχουν μια διεθνή διάσταση για το TTIP. Και για το τι μπορούμε να πετύχουμε. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Δεν διαπραγματευόμαστε τα πρότυπα δεν είναι διαπραγματεύσιμα. Δεν είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε τα πρότυπα ασφάλειας των τροφίμων. Είπατε ότι και οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, θα πρέπει να μπορούν να δεχτούν την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Για μας είναι θεμελιώδους σημασία. Πρέπει να μας δεχτούν ως σύνολο και όχι να ασχολούνται ή να ασχολούμαστε εμείς με αναχώρα προσεγγίσεις, δηλαδή διμερός. Αυτό θα κατέστρεφε την εσωτερική μας αγορά και την κοινή γεωργική μας πολιτική, καθώς και τα κοινά μας πρότυπα. Και από την πλευρά μας, μιλώντας για υγειονομικά και φυτο μέτρα, Προφανώς προτιμούμε να έχουμε υψηλά πρότυπα και να στέλνουμε στις ΗΠΑ σαφή μηνύματα ότι τα πρότυπά μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά είναι, είναι τα θεμέλια επί των οποίων θα συνεχίσουμε και θα οικοδομήσουμε το διάλογό μας. Σε ό,τι αφορά το αναπαραγωγικό υλικό των φυτών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όντω απέσυρε τον Φεβράριο του 2015 την πρότασή τη για το θέμα αυτό. Διότι κάποια θέματα της προτινόμενη νομοθεσίας εντοπίστηκαν από την αξιολόγηση ήδη που είχε γίνει το 2007-2008 όμως οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις εντόπισαν κάποια σημεία προβληματικά. Τους τελευταίους μήνες λοιπόν συνείδησα όλους τους εκπροσώπους των κυβερνητικών οργανώσεων που μας πρότειναν νέες προσεγγίσεις για το θέμα αυτό. Όμως σήμερα μας ενδιαφέρει να συζητήσουμε με όλους τους ενδιαφερομένους τον τρόπο που θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Υπάρχουν δύο επιλογές. Η μία είναι να ανανεώσουμε την προηγούμενη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κάποια άρθρα να αλλάξουν με την επιλογή να αξιολογήσουμε ή να έχουμε μία ε, εν μέρη αξιολόγηση αντικτύπου για τα θέματα αυτά ή να προβλέψουμε μια νέα προσέγγιση, τελείως νέα, η οποία θα μας επιτρέπει να ξεκινήσουμε αυτή τη νέα μελέτη αντικτύπου. Όμως θα χρειαστεί χρόνος, τουλάχιστον δυόμιση χρόνια. Σε ό,τι αφορά το γλυφοζάντ. Στο κατά το Σαββατοκύριακο είχαμε μία καταγγελία από τον Διεθνή Οργανισμό κατά του Καρκίνου για να, το για να καταγράψουμε αυτή την ουσία στον κατάλογο των καρκινογόνων ουσιών. Το γλυφοζάντ είναι ένα συστατικό κάποιων γενετικώς τροποποιημένων ε, καλλιεργιών. Και η έγκριση που έχει δοθεί εδώ ε, σε κάποια ζυζανιοκτώνα λέγεται την 31η Δεκεμβρίου 2015. Και αυτή η διαδικασία αναθεώρησης ε, πάντοτε ε, ισχύει στην περίπτωση εκπνοής της άδειας κάποιων ζυζανιοκτώνων. Ούτως ή άλλως τρέχει λοιπόν φέτος η Γερμανία και κάποια άλλα κατημέλη βάσει διεξοδικών επιστημονικών στοιχείων λένε ότι η ουσία αυτή δεν είναι ανάγκη να καταγραφεί και να ενταχθεί μεταξύ των καρκινογόνων. Αργότερα το 2015 θα υπάρξει μια γενικότερη αξιολόγηση για την ισχύουσα νομοθεσία. Και για τα νοικοτινοειδή. Δεν προβλέπεται εδώ μελέτη αντικτύπου. Η ΕΦΣΑ έχει ξεκινήσει μια διαδικασία ανοιχτή για την υποβολή δεδομένων. Μόνο στο τέλος της διαδικασίας αυτής μελέτης θα αποφασίσουμε τα επόμενα βήματα. Uh, about Και μιλώντας για την ε, ζωή των ζώων και τα αντιβιωτικά. Κάποια πράγματα μπορούν να επιτευχθούν σε εθνικό επίπεδο. Ο ίδιος εγώ επισκέφθη ένα σύγχρονο αγρόκτημα στις κάτω χώρες ε, που ασχολείται ακριβώς με τον περιορισμό χρήσης αντιβιωτικών. Τέτοια είναι τα παραδείγματα που θέλουμε να λάμψουν και να φωτίσουν τους υπόλοιπους. Βεβαίως, Ευχαριστώ να απαντήσω και στις ερωτήσεις σας γραπτός. Είναι μεταξύ των υποχρεώσεών μου. Ευχαριστώ πολύ. Και ζητώ συγγνώμη κύριε Επιτροπή, απαντήσατε σε πολύ μεγάλο βαθμό λεπτομέρειες ερωτήσεις που σας ε, ετέθησαν. Εάν βεβαίω χρειαστεί να δώσετε πιο πολλές ε, λεπτομέρειες, ασφαλώς μπορείτε και γραπτός να συνεχίσετε την επικοινωνία με τους συναδέλφους και όλοι βέβαια γνωρίζουμε ότι ένα πάσα στιγμή μπορούμε να απευθύνουμε ερωτήσεις στον Επίτροπο. Καθώς ο δε μάλλον ο Επίτροπός μας πάντα είναι διαθέσιμος να απαντήσει στις ε, προτάσεις και τα αιτήματά μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Δείξατε μια σειρά από θέματα, τις διάφορες απειλές που μας ε, απασχολούν τις ασθένειες στην Ανατολική και την Νότια Ευρώπη, τις διαπραγματεύσεις. Πολλά θέματα έχουμε να συζητήσουμε κύριε Επίτροπε και ελπίζουμε ότι ο διάλογος αυτός θα παραμείνει ενεργός. Ολοκληρώνουμε λοιπόν αυτό το πρώτο σημείο και σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Αλλά θα διακόψουμε πρώτα για να το χαιρετήσουμε τον Επίτροπο. Και τώρα περάμε στο σημείο 5. Παρουσίαση από την Επιτροπή. Όχι, λέει πρόεδρος, το συγγνώμη. Η κυρία Νότλιχ είστε στο λόγο, παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Μια μικρή διακοπή είπα. Συνεχίζουμε τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Είχα κάτι να σας παρακαλέσω. Εσάς και την κυρία και στην κερδικά ε, που έχει τη σχετική εισήγηση. Είμαι σκιώδης ηγήτρια στο θέμα της κυρίας Κιώστιγκερ και βλέπω ότι για τη νέα δασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουμε να ψηφίσουμε αύριο ε, έχουν κατεθεί πολλές τροπολογίες. Πρέπει να τα συνεννοηθούμε όλα αυτά. Παρακαλώ λοιπόν την κυρία Κιούστιγκερ να ε, μας πει αν μπορούμε να κάνουμε την ψηφοφορία την Πέμπτη και εσείς βέβαια να μας πείτε γιατί είναι πολύ μεγάλη πίεση του χρόνου. Αν μπορέσουμε να αναβάλουμε θα έχω την ευκαιρία να προετοιμαστώ καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάνι ε, Κυρία Νόχτλ, ξέρετε ότι δεν μπορώ να πάρω μόνο μου αυτή την απόφαση. Πρέπει να τηρήσουμε κάποιες διαδικασίες. Ερωτώ αν υπάρχουν τουλάχιστον δύο βουλευτές που ε, δέχονται και υποστηρίζουν την πρόταση της συναδέλφου. Παρακαλώ να εκδηλώσουν την υποστήριξή τους. Μάλιστα, πολύ ωραία, δύο άτομα τουλάχιστον από ό,τι βλέπω. Τέσσερι βουλευτές υποστηρίζουν το αίτημα. Μάλιστα. Οι συντονιστέ τι μα λένε. Πρέπει να συμφωνούν και οι συντονιστέ. Υπάρχουν αντιρρήσει. η κυρία Κώστην και στην καιρό συγκεντρία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με εξαφνιάζει το ότι η κυρία Νόιχλ δεν έχει προλάβει να ετοιμαστεί να κοιτάξουμε λίγο την ιστορία αυτού του θέματος, τη στρατηγική για τα βάση. Την έχει καταθέσει Σεπτέμβριο του 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην προηγούμενη θητεία του το Κοινοβούλιο είχε και αυτό έκθεση πρωτοβουλίες, ε, πρωτοβουλίας. Πάλι δεν είχε προλάβει να ολοκληρώσει. Σεπτέμβριο πέρσι ξεκινήσαμε την επεξεργασία της έκθεσης ε, με 460 τροπολογίες όντως. Αλλά θέλω να λάβετε και υπόψη ότι πρόκειται για μια έκθεση πρωτοβουλίας και όχι για νομοθετική πράξη η σκιώδη συγκεκριά των σοσιαλιστών εξ αρχής ε, έχει εμπλακεί στη δικασία ε, βεβαίως να μην μπόρεσε να είναι πάντα παρούσα. Πάντως μπορέσαμε να διατυπώσουμε 29 συμβαστικέ τροπολογίες και νομίζω ότι αυτές για μια έκθεση πρωτοβουλίας είναι αξιόλογο νούμερο. Ε, πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε την ψηφοφορία αύριο. Είχαμε μέχρι την προηγούμενη Παρασκευή το χρόνο για την κατάθεση τροπολογιών ως προς τον κατάλογο των ψηφοφοριών. Έχουν καταθέσει σχετικά 20 τροπολογίες σοσιαλιστές. Προσπαθήσαμε να κάνουμε δεκτές και να εντάξουμε στον κατάλογο τις προτάσεις του στο μέγιστο δυνατό βαθμό, όσο και αν οι δημοκρατικές διαδικασίες δεν επιτρέπουν πάντοτε να γίνονται δεκτά όλα τα αιτήματα του ενός, αλλά νομίζω ότι τους έχουμε ικανοποιήσει σε μεγάλο βαθμό. Και εν πάση περιπτώσει δεν νομίζω ότι αυτό έχει τόσο μεγάλη σημασία σε σχέση με τη γνώμη που θα δημοφώσει το Κοινοβούλιο. Παρακαλώ να έρθουν αύριο οι συνάδελφοι για την ψηφοφορία. Έχουμε χάσει αρκετό χρόνο όπως είπα και με όλη ε, την εκτίμηση που έχω για, την, ε, για τις επιφυλάξεις συναδέλφου. Η Γραμματεία έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να οργανώσει τα πάντα, να συνδυάσει όλους τους ε, παρισταμένους και γι' αυτό καλό είναι να μην καθυστερήσουμε παραπάνω με την ψηφοφορία και να μπορέσει να πάει το θέμα στο ε, Στρασβούργο, στην Ολομέλεια και να προσδοριστεί η στρατηγική του Κοινοβουλίου. Ο πρόεδρος ευχαριστώ. Χωρίς να θέλω να κάνω μεγάλο διάλογο θα πάρει το λόγο η κυρία Μίλλερ τώρα. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστώ την κυρία και Κέστιγκερ για την εξαίρετη επεξεργασία της εκθέσεως και το έγγραφο που είχαμε που ήταν εξαίρετο και πολύ καλά ισορροπημένο. Την τελευταία, τις τελευταίες εβδομάδες το επεξεργαστήκαμε εντατικά. Καταλήξαμε σε μια καλή συμβαστική ε, λύση. Συναντηθήκαμε επανειλημμένως, επεξεργαστήκαμε εντατικά τις προτάσεις. Αυτό που μας λέγεται τώρα, αυτό που μας έχει υποβληθεί τώρα είναι ένα κείμενο περιεκτικό και ισορροπημένο ε, θα παρακαλέσω λοιπόν να μην αποσυρθεί, να προχωρήσουμε αύριο στην ψηφοφορία. Είμαστε έτοιμοι. Όλοι έχουμε δουλέψει πάνω στο έγγραφο, έχουμε κάνει πολλούς συμβασμούς και πολλά πράγματα τα οποία εγώ δεν είχα πολύ όρεξη να καταπιώ, τα κατάπια. Γι' αυτό λοιπόν έχει έρθει πια η ώρα να ψηφίσουμε. Ο Πρόεδρος. Λοιπόν, κοιτάξτε. Αύριο θα γίνει και η συζήτηση με τον Επιτροπό Χόγκαν. Με την ευκαιρία αυτή θα είμαστε όλοι παρόντες. Άρα μπορούμε πριν ακριβώς από αυτό, πριν από τη συζήτηση με τον Επίτροπο, να κάνουμε την ψηφοφορία. Κυρία Κιώστιγκερ, ναι, μια ερώτηση προς την κυρία Μιλόρ δικαστικά. Μπορούμε δηλαδή να πάσα στιγμή σε μια συνεδρίαση να καταθέσουμε το αίτημα για την αναβολή ενός θέματος. Γιατί το γνωρίζαμε εδώ και καιρό ότι επρόκειτο να γίνει η ψηφοφορία. Από την αρχή όλοι έχουν ε, συμφωνήσει, έχουν συνεργαστεί, έχουν οριστεί τροπολογίες, έχουν καταθέσει προτάσεις. Δεν βλέπω λοιπόν γιατί δεν πρέπει τώρα να ψηφίσουμε. Όλοι έχουμε τηρήσει τι προθεσμίε μα, έχουμε κάνει ο καθένα το μερίδιο από τη δουλειά του. Η δουλειά, δουλειά τη γραμματεία ήταν επίση εξαίρετη, το είπα νωρίτερα. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι στον κατάλογο των τροπολογιών που θα μπορούσε να αλλάξει μέχρι την Πέμπτη. Δεν βλέπω, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει τώρα να διευκρινίζουμε ή να ε, ρυθμίζουμε, διευθυντούμε ζητήματα της δημοκρατίας τώρα με έναν τέτοιο τρόπο. Νομίζω ότι πρέπει να ψηφίσουμε αύριο ο Πρόεδρος. Αν θέλει η Γραμματεία σύντομα να μας ενημερώσει για τη διαδικασία. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Για να απαντήσω στην κυρία Κίστιγκερ, όντω το άρθρο 194 παράγραφο του κανονισμού επιτρέπει στον κάθε βουλευτή να ζητήσει την αναβολή ψηφοφορία πριν από την έναρξη των ψηφοφοριών, αναλογικά των διατάξεων που ισχύουν για τι ψηφοφορίε στην Ολομέλεια και εφόσον υποστηρίζουν τρει βουλευτέ τουλάχιστον το αίτημα, μπορεί αυτό να αποφασιστεί. Αφού δεν υπάρχει όμω συνένεση, θα πρέπει να γίνει ψηφοφορία για το αν θα γίνει η ψηφοφορία όπω προβλεπόταν, όπω πρότεινε ο πρόεδρο, δηλαδή αύριο το πρωί, να ψηφίσουμε εάν ή όχι θα ε, παραμείνει στην εμερήσια διάταξη για τις 3 το απόγευμα η ψηφοφορία για την ε, δασική στρατηγική ο Πρόεδρος. Καλώς. Δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο. Κύριε Νόχιλ, όχι. Πολύ καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Ακούσαμε τις διαφορετικές τοποθετήσεις. Και προχωρώ. Σημείο 5. Παρουσίαση από την Επιτροπή σχετικά με την κλεψιέλα και παρακαλώ τον εκπρόσωπο της Επιτροπής να λάβει το λόγο. Αλλά Παρακαλώ, να είστε όσο δυνατόν πιο σύντομοι. Πολλές πληροφορίες ήδη τις λάβαμε. Μας έδωσε και ο Επίτροπος μια ενημέρωση. Παρακαλώ λοιπόν να γίνει πολύ σύντομα η ενημέρωση πλευράς της Επιτροπής. Ποιος είναι εδώ από την Επιτροπή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να στήσω συγγνώμη που επαναφέρω το θέμα αυτής της ε, κλεψιέλας, αλλά έχω και κάποιες εικόνες να σας δείξω για τη ζημιά μπορεί να προκαλέσει. Για πρώτη φορά εμφανίστηκε στην Ευρώπη η ασθένεια αυτή που πλήττει ελαιόδαντρα στην Νότια Ιταλία και κυρίως στην περιοχή της Πούλια μας έχει ενημερώσει από τον Οκτώβριο του 2013 η Ιταλική κυβέρνηση για, την πρώτη, για το πρώτο κρύγουρσμα που ανοιχνεύτηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λάβαμε το 2013 σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέτρα κατεπήγοντα, τα οποία καταγράφηκαν με πιο λεπτομερή τρόπο τον Ιούλιο του 2014 σε ένα έγγραφο με τα οποία μέτρα ορίζουμε πολύ αυστηρές προδιαγραφές για την εισαγωγή και τη διακίνηση αυτών των φυτών, έλεγχος ε, στις πληγήσεις περιοχές και εκρίζωση όλων των ε, στενών δέντρων, ελαιοδέντρων συγκεκριμένα και αυτό βάσει και των δηλώσεων που είχαμε λάβει από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Έκτοτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πραγματοποιήσει δύο ελέγχους από την Υπηρεσία τροφίμων και κτηνιατρικής ε, το 2014, το 2 το Νοέμβριο του 2014, που δυστυχώς διαπίστωσαν ότι έχει επιδεινωθεί σημαντικά η κατάσταση μετά τον πρώτο έλεγχο του Φεβρουαρίου του 2014. Επίσης, τα μέτρα μας από αποσκοπούν στην εκκριζωσή της ασθένειας καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι επικεντρώνονται μόνο στον περιορισμό οι δράσει των αρμοδίων αρχών και όχι στην εκκρίζωση τελείως της ασθένειας. Είναι πολύ περιορισμένο ο αριθμός των ελαιοδέντρων που έχουμε μέχρι τώρα εκκριζωθεί ή αφαιρεθεί. Δυστυχώς η Ιταλία πρόσφατα μας ενημέρωσε για ακόμη ένα κρούσμα εκτός της περιοχής όπου πρώτα εντοπίστηκε η νόσος και που είχε ήδη περιχαράξει η Ιταλία. Στο Μπρίντιζι βλέπουμε ε, τα νέα κρούσματα στην περιοχή του Μπρίντιζι, δηλαδή κινείται πλέον η ασθένεια έξω από την αρχικά σε περιοχή. στην αρχική δήλωση του 2013 για τα διάφορα μέσα, την αρχική μάλλον ακολούθησε μια άλλη της ε, Υπηρεσίας Φαρμακών και Υγείας για του 2015 για τον κίνδυνο που μπορούσαν ε, να σημάνουν ε, κρούσματα τέτοιου τύπου για τα εσπυριδοειδή και τα κλίματα. 200 διαφορετικά είδη, πολύ περισσότερα δηλαδή από όσα καλύπτουν τα ισχύοντα μέτρα. Η ασθένεια δεν έχει εμφανιστεί ακόμη σε ευρωπαϊκό έδαφος σε σπυριδοειδή και κλίματα και η έκταση των φυτών αυτών ε, που, ερευνούνται για αυτή την νόσο στην Πούλια είναι όλο και μεγαλύτερη γιατί προχωρούν οι έλεγχοι. Ανακοινώνονται λοιπόν μια σειρά από έλεγχοι από τις Ιταλικές Αρχές με σημαντική και οικονομική υποστήριξη. Από τα αποτελέσματα όμως που βλέπουμε σχέση με την εξέλιξη της νόσου, διερωτώμεθα αν θα αρκέσουν αυτά για να παρεμποδίσουν την περαιτέρω διάδοση της ασθένειας. Υπάρχουν επαφές διαρκείς με τις τελικές αρχές προκειμένου να βρούμε την καλύτερη λύση. Είχαμε σε ανώτερο επίπεδο τρεις συνεδριά την προηγούμενη εβδομάδα με τις τελικές αρχές. από τα νέα ευρήματα και την γνωμοδότηση του ΕΦΣΑ προχωρεί η αξιολόγηση των κατεπηγόντων μέτρων μας. Σας διαβεβαιώ ότι ο κατάλογος των φυτών που ενδέχεται να ε, νοσήσουν έχει διευρυνθεί ακόμη περισσότερο από την έκθεση του ΕΦΣΑ. Ο κατάλογος αυτός θα πρέπει να καλύψει όλα εκείνα όλους εκείνους πιθανούς κινδύνους και προσπαθούμε να ενισχύσουμε τους περιορισμούς ε, για τη, στην κίνηση έξω από, τους, ε, από, έξω περιοχές που έχουν πληγεί και τις χώρες που έχουν πληγεί με πολύ μεγάλη προσοχή. Προβλέπετε, για να σας ενημερώσω, να γίνει τεχνικού επίπεδου ανταλλαγή απόψεων με τα κράτη-μέλη μέχρι το τέλος της εβδομάδας Ανάλογα δε με την έκβαση αυτών των συνομολιών ε, και βέβαια των εργασιών σε επίπεδο επιτροπής, αναμένεται ψηφοφορία για την περαιτέρω ενίσχυση των, μέτρο, μέτρων από την μόνιμη επιτροπή τον Απρίλιο. Μια σειρά από ζητήματα εγέρθησαν σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που για λόγους χρόνου δεν μπορέσαμε να απαντήσουμε. Έχουν να κάνουν με την έρευνα ορισμένα, ο Επίτροπος Ανδρουκαίτης είναι σε επαφή με τον Επίτροπο για την Γεωργία και την Έρευνα και ζητάει να μπει η κλεψιέλα σε πιο υψηλό ε, επίπεδο προτεραιότητας από τον κατάλογο ε, για την έρευνα, πράγμα το οποίο μάλλον θα επιβεβαιωθεί αλλά δεν το έχουμε ακόμα την επιβεβαίωση, για τις αποζημιώσεις υπήρξε ένα ζήτημα, ένα ερώτημα. Η νομοθεσία μας μέχρι σήμερα δεν επιτρέπει την αποζημίωση του γεωργού πέραν των δαπανών που έχουν να κάνουν με την εκρίζωση του φυτού, του δέντρου. Δεν έχουμε δηλαδή δημοσιονομικά μέσα με βάση την ισχύουσα νομοθεσία του κανονισμό μας για να ε, αποζημιώσουμε για μακροπρόθεσμη οικονομική απώλεια εσόδων στο χώρο της γεωργίας. Αυτά και αν υπάρχουν ερωτήσει, πολύ ευχαριστώ να απαντήσω. Σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Έχουν ζητήσει αρκετοί το λόγο. Θα ήθελα να σας ζητήσω παρακαλώ να είστε σύντομοι. Η κυρία Ράντς Γκαρσία. Σας ευχαριστώ. Έχει τεθεί το θέμα της ξυλέλια φαστιντιόζα από το 2012 και υπάρχει τεράστια ανησυχία από πλευράς των ελαιοπαραγωγών. Πριν λίγο καιρό είχα συναντηθεί στην Κόρδοβα σε μια συνάντηση ε, των ελαιοπαραγωγών με εμπειρογνώμονες από την Ευρώπη και η ανησυχία τους είναι τεράστια. Είναι τεκμηριωμένη για αυτό το βακτήριο το οποίο δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην Ιταλία αλλά απειλεί το σύνολο της Μεσογειακής Λεκάνης. Το πρόβλημα παραμένει το 2015 δεν έχουμε όμως συζητήσει το θέμα όσο ε, του αξίζει θα έλεγα. Οι συνέπειες είναι τεράστιες. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο να αντιμετωπίσουμε. Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι τα μέτρα τα οποία ε, θα εφαρμόσει το Ιταλικό κράτος δεν επαρκούν. Ε, επίσης έχουμε το πρόβλημα της εισαγωγής ε, δένδρυλίων ε, και φυτών γενικότερα από χώρες στις οποίες υπάρχει η ασθένεια αυτή, σοβεί η συγκεκριμένη αυτή ασθένεια. Λοιπόν θα πρέπει να αποφύγουμε τέτοιου είδους καταστάσεις και να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι θα κάνει έτσι ώστε αυτή η ασθένεια να θίξει το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το σύνολο της Μεσογειακής περιοχής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Αντριέ. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας της φυτικής παραγωγής και τίθεται το θέμα των φυτών που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έθεσε και ο Ανδρουκάητης ο Επίτροπος. Δεν είναι κάτι το καινούριο, το συζητήσαμε και κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περίοδου. Στα πλαίσια των συζητήσεων οι οποίες έγιναν είχα εκφράσει τις ανησυχίες μου για τις ελλείψεις της στρατηγικής ελέγχου η οποία δεν μας προστατεύει και το βλέπουμε σήμερα, δεν προστατεύει επαρκώς το κοινοτικό έδαφος από την είσοδο βλαβερών οργανισμών. Και παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλει να τροποποιήσει το υπάρχον σύστημα. Εγώ στα πλαίσια της συζήτησης που είχε γίνει είχα πει να υπάρξει μια νέα στρατηγική ελέγχου η οποία να βασίζεται στην διαχείριση των κινδύνων, συμβατών κινδύνων με αυτούς που περιλαμβάνουν οι διεθνείς συμβάσεις ε, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Έχω λοιπόν δύο ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άκουσα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αρχίσει να σκέπτεται κάποια μέτρα, αλλά μήπως θα πρέπει να αλλάξει τη στρατηγική ελέγχου την οποία χρησιμοποιεί. Και υπάρχει και το θέμα των αποζημιώσεων. Πώς πιστεύει ότι θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες αυτού του βακτηρίου, το οποίο δυστυχώς θα προστεθεί και σε άλλα παράσιτα, όπως... Ε, Donc, euh, et parce que les solutions techniques de lutte en raison de la non-autorisation τις λιχίνες οι οποίες προσκολώνται στα ελαιόδενδρα ε, και δυστυχώς ο συνδυασμός των δύο μπορεί να αποβεί ιδιαίτερος επικίνδυνος. Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λέει ο κ. Νταντά. Ε, άκουσα ότι ορισμένα εδάφη της περιφέρειάς μου θίγονται, όχι σε επίπεδο ελαιοδένδρων, αλλά αυτό το βακτήριο φαίνεται ότι περνάει και στην αμπελοϊνική παραγωγή όπως επίσης και στα εσπεριδοειδή. Désormais en Corse, alors les Το ερώτημά μου λοιπόν αναφέρεται στην ταχύτητα απάντησης, αν θέλετε, ε, ανταπόκρισης ε, σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Αυτό το οποίο μετράει σε τέτοιου είδους καταστάσεις είναι η ταχύτητα απόκρισης. Έχετε λοιπόν ένα χρονολόγιο αντίδρασης μπροστά σας. Eh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αναφέρθηκε σε αυτά τα οποία συζητήθηκαν στην Κόρδοβα η συνάδελφο Σαράντσα. Εγώ είμαι από την Ανδαλουσία, η οποία είναι μια πλούσια περιοχή σε ε, ε, ε, ελαιοπαραγωγός περιοχή και έχει μεγάλη σημασία αυτή η καλλιέργεια. Μας απασχολεί ιδιαιτέρως η κατάσταση αυτή που έχει δημιουργηθεί θεωρούμε ότι δεν υπάρχει ένας ουσιαστικός έλεγχος και ακριβώς γι' αυτό υπάρχουν πάρα πολλές ανησυχίες σε περιοχές όπως η δική μου αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές περιοχές. Γιατί επαναλαμβάνω ότι τα μέτρα τα οποία έχουν λάβει μέχρι τώρα είναι γενικά ανεπαρκή. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν τι θα γίνει από εδώ και πέρα, τι μέτρα τα οποία θα πάρετε έτσι ώστε να υπάρχει εισαγωγή αντίστοιχων μολυμένων φυτών. Από μεγάλους λιμένες ε, πώς θα υπάρξει καλύτερος έλεγχος ιδιαίτερα σε μεγάλους επαναλαμβάνω λιμένες ε, εισαγωγής φυτικών ε, ουσιών, φυτικών προϊόντων. Ε, θα υπάρξει μια αντιμετώπιση του μολυσμένου φυτικού υλικού για να αποφύγουμε τέτοιες καταστάσεις και σε άλλες χώρες. Ο κύριος Καπούτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κλεψιέλα καταστρέφει ολόκληρη περιοχή στην Ιταλία, ιδίως στην Απουλία. Ολόκληρες εκτάσεις. Άκουσα τι είπε η Επιτροπή και βλέπω ότι χρειάζεται εδώ ιδιαίτερο συντονισμός με όλα τα κράτη-μέλη. Ο διακρατικός συντονισμός είναι απαραίτητος. Η Ιταλία και η Επιτροπή ακόμη δεν έχουν την απαραίτητη μορφή συνεργασίας από ό,τι φαίνεται, όπως είπε και ο κ. Σαντιουκάτης. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ε, η φάση του ελέγχου, το στάδιο του ελέγχου. Και θα συμφωνήσω με τον συνάνδρεφο Άγγλιο ότι πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία λήψη αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το είχα πει και με άλλη ευκαιρία ενώ ε, ο γιατρός ε, ξεφυλίζει τον χειρίδιο μπορεί ο ασθενής να εκπνεύσει. Ε, εδώ λοιπόν μιλάμε για μια γεωργική παραγωγή πολύ σημαντική για την Νότια Μεσόγειο. Και ό,τι διαφωνίες και αν υπάρχουν, σίγουρα η νομοθεσία πρέπει να προσαρμοστεί μακροπρόθεσμα, αλλά και τώρα πρέπει να βιαστούμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη, διότι θα πρέπει να μακρηγορήσω γιατί έρχομαι από την Απουλία, από το Σαλέντο συγκεκριμένα. Και πρέπει να διευκρινίσω ότι εδώ για μια ουσιαστική ε, ταχεία ξύρανση της ελιάς. Δεν είναι απλώς μια αρρώστια του ξύλου. Την ε, περασμένη εβδομάδα ο Επίτροπος Φιλέτη, για, που είναι ο Επίτροπος της Ιταλικής Κυβέρνησης για να αντιμετωπίσει αυτή την κατεπίγουσα ανάγκη, ε, με 13 εκατομμύρια ευρώ πρόκειται να εκριζώσει με ειδικά εργαλεία τα άρρωστα δέντρα και με στις 30 Μαΐου θα γίνει αυτό για, τις, για τα ελαιόδεντρα και στις 30 Ιουλίου για τα ποροφόρα. Ε, όλα αυτά με χημικές ουσίες και εκρίζωση σε ολόκληρη την γεωγραφική αυτή ζώνη. Είναι τεράστια, εκτεταμένη 50 επί 15 χιλιόμετρα και οι άλλες περιοχές και οι περιοχές με κρίσιμα κρούσματα. Το πρόγραμμα θα αποφασιστεί στις 26-27 Μαρτίου στα πλαίσια της Μονίμης Επιτροπής για την Υγεία των Φυτών. Εδώ έχουμε όμως επιστημονικές αμφιβολίες. Δεν αποδεικνύεται ότι το βακτήριο Λεψιέλα είναι η μόνη αιτία της ασθένειας. Οπότε όλο αυτό, ε, ακριβώς αυτό που ζητούμε είναι βάσει συγκεκριμένων αποδεκτικών στοιχείων, βάσει των γεωπόνων που έστειλε στο Σαλέντο ήδη από το Φεβρουάριο η Επιτροπή να μας ενημερώσει για τον ε, έλεγχο που έγινε. Με συγχωρείτε αλλά είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν ε, μελέτες της ΕΦΣΑ και της DG που δείχνουν ότι η κρίζωση δεν είναι η καλύτερη λύση και επειδή βλέπω ότι σηκώνεται το σφυρί πρόεδρε, ε, να σας παρακαλέσω να μελετήσετε πολύ καλά την κατάσταση. Υπάρχουν και μήκητες, υπάρχουν και άλλα παθογόνοι παράγοντες. Εδώ πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτό μπορεί να αφορά όλη την Ευρώπη, όχι μόνο την Απουλία. Και πρέπει κυρίως να καταλάβουμε γιατί... Ε, παρά ε, την, την εισαγγελία και την ε, παραγγελία για έρευνα που είχε κάνει, να μην ξεχνάμε ότι απαιτείται επιστημονική τεκμηρίωση. Είναι σαν να θέλουμε να θεραπεύσουμε το AIDS, σαν να επρόκειτο για πνευμονία. Πρέπει λοιπόν εδώ να είμαστε αυστηρότατοι στα επιστημονικά στοιχεία στα οποία βασιζόμαστε να δούμε ποια είναι η αιτία, η γενεσιουργός αιτία και να αντιληφθούμε ότι η κατάσταση ναι είναι κρίσιμη αλλά το Ιταλικό κράτος δεν λαμβάνει τα σωστά μέτρα και μάλιστα με επιστημονικές αποδείξεις. Ζητούμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει την κατάσταση και να γίνουν μελέτες για την επίπεδο ε, με πανεπιστημιακή συμμετοχή και ε, ρωτώντας τους παραγωγούς που ξέρουν τι πρέπει να κάνουν για τα δέντρα τους. Rozumiemy Pani sytuację, Καταλαβαίνω πολύ καλά την κατάσταση. Ζητάτε περισσότερο χρόνο αγόρευσης μεν, αλλά καλό είναι τις πληροφορίες να μπορείτε να τις αναφέρετε και στην Επιτροπή για να ενισχυθούν τα επιχειρηματά σας. Μιλάμε για μία μάστιγα η οποία έχει καταστρέψει χιλιάδες δέντρα στο νότο της Ιταλίας. Η μάστιγα αυτή αποδεικνύει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών μπορεί να είναι καταστροφική. Βλέπουμε ότι κάποια φυτά τα οποία εισήχθησαν από την Κοσταρίκα ε, προκάλεσαν την καταστροφή αυτή. Ε, επίσης μπορεί να χτυπήσει και το αμπέλι γιατί ταλαιπώρησε πολύ το αμπέλια στην Καλιφόρνια. Είναι αδύνατο να αντιμετωπιστεί η μάστιγα αυτή και δεν υπάρχει προς το παρόν αντίδοτο. Νομίζω λοιπόν ότι σήμερα ε, είναι απαραίτητο να απαγορεύσουμε την εισαγωγή ε, φυτικών εν ζωή προϊόντων από άλλες χώρες, από τη Βόρειο Αφρική και να υπάρξει απαγόρευση ιδίω εισαγωγή αμπελιών και ελαιοδένδρων από άλλες χώρες. Ο κύριος Ταραμπέλα. Ευχαριστώ. Μετά από τους προλαλήσαντες φυσικά εγώ θα ε, ταχθώ με αυτούς οι οποίοι ζητούν ε, μεγαλύτερες ε, επιστημονικές αποδείξεις. Η κυρία Νταμάτο μίλησε με πάθον γιατί μιλάμε για την απουλία, για δέντρα τα οποία έχουν εκατοντάδες χρόνια ζωής και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να, πάρουμε, να, να λάβουμε τα πολύ σημαντικά μέτρα Άκουσα για, για διακοσμητικά φυτά που εισάγονται από την Κωνσταντίνα. Άκουσα για φυτά καφέ τα οποία εισάγουμε από τη χώρα αυτή. Πρέπει να σταματήσουμε τις εισαγωγές. Είναι ξεκάθαρο. Πρέπει να συνδυαστούν οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι προσπάθειες της Ιταλίας. Και ίσως θα είναι απαραίτητο σε τέτοιου είδους κρίσεις να υπάρξει ένα σύστημα σαν και αυτό Έχουμε το Rapid Exchange, το RAPEX για τους καταναλωτές. Ε, εγώ συμφωνώ ότι αυτό το οποίο χαρακτηρίζει την αντίδρασή μας είναι ο αργός, ο αργός χαρακτήρας. Τώρα για τα ζωτούχα ίσως θα πρέπει να επιτρέψουμε κάποια απαγορευμένα φάρμακα μόνο και μόνο για να σταματήσουμε την επέκταση της ασθένειας. Ίσως λοιπόν απαιτούνται περισσότερα και πιο επίγοντα μέτρα. Ευχαριστώ. Πράγματι δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να προσαρμόσουμε την ομοθεσία μας σε τέτοιου είδους καταστάσεις για να προετοιμάσουμε τα προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν στο μέλλον. Οι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής έχουν το λόγο για να δώσουν απαντήσεις. Παρακαλώ λίγο σύντομα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόεδρε, ακούστηκαν διάφορες διαφορετικές απόψεις. Άλλοι ζητούν να πάμε πολύ γρήγορα, άλλοι μας ζητούν να εξετάσουμε προσεκτικά όλες τις επιστημονικές ε, μελέτες. Να ξεκινήσω από εκεί λοιπόν. Μας ε, πλησιάζουν διάφορες οργανώσεις σχετικά με την, με την πληροφορία ότι αυτά δεν οφείλονται, αυτές οι άρρωσες δεν οφείλονται στην κλεψία, αλλά σε μήκητα. Κοιτάξτε, είμαστε σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές, ζητούμε την αξιολόγηση από τις αρμόδιες αρχές, από τον ΕΦΣΑ, που, είναι τα, που έχει τα ορόσημα τα επιστημονικά, να μελετήσουν τα στοιχεία και θα θέλαμε να έχουμε μια σαφή δήλωση και τοποθέτηση που να επιβεβαιώνει ή να διαψεύδει τις πληροφορίες σχετικέ με την κλεψίαλα πριν να λάβουμε αποφάσεις για οριστική δράση. Για τα άλλα ζητήματα, σαφές χρονοδιάγραμμα, για το πότε θα αντιδράσουμε, όπως είπα και νωρίτερα θα έχουμε μια πρώτη αρχική συζήτηση με τα κράτη-μέλη και τη Ρυθμιστική Επιτροπή με βάση τη συζήτηση αυτή και την παρακολούθηση, την συνέχεια που θα δοθεί στην αρχική συζήτηση μεταξύ Επιτροπής και Τελικών Αρχών θα υιοθετηθούν νέα μέτρα μέχρι τα Απριλίου, όπως είπα. Κάποια σημεία επίσης που αναφέρθηκαν σχετικά με τα μέτρα που θα ληφθούν στο μέλλον. Είπα στην παρέμβασή μου στην αρχή ότι θα ενισχυθούν τα μέτρα και ότι θα ενισχυθεί σημαντικά, θα διευρυνθεί σημαντικά ο χώρος, η περιοχή που καλύπτεται ε, από την υποχρέωση τήρηση των φυτογειονομικών μέσων, που τώρα είναι μόνο η πουλή της Ιταλίας. Μάλλον το Λέτσε, και θα επεκταθούν τα μέτρα και σε άλλες περιοχές. Και να διορθώσω εδώ το εξή ε, που ακούστηκε ότι δεν έχει πει η Επιτροπή ότι, ή, ότι δεν είναι δυνατόν να εκριζωθεί η ε, νόσος, αλλά ότι σε αυτό το στάδιο δεν είναι πλέον δυνατόν. Δηλαδή προσπαθούμε να συγκρατήσουμε και να εμποδίσουμε την διαδοσή της άλλες περιοχές, είτε της Ιταλίας, είτε της Μεσογείου, είτε και άλλων κρατών μελών ανάλογα με τα είδη τα καλλιεργούμενα. Έχουμε μέτρα παραδείγματι που προτείνουν πολύ μεγαλύτερη ζώνη ασφαλείας και υποχρέωση εκρίζωσης ε, των ε, νοσούντων δέντρων και για τις περιοχές που γειτονεύουν με την, αυστηρή, με την ε, εκτεταμένη αυτή ζώνη ασφαλείας. Αλλά όλα αυτά θα γίνουν σε συζήτηση με τα κράτη-μέλη και κυρίως με την Ιταλία που σε τελευταία ανάλυση είναι η αρμόδια, περισσότερο αρμόδια για να αντιμετωπίσει τα ζητήματα. Επίσης πρέπει να γίνει ένα, να επιβληθεί ένα πιο αυστηρό καθεστώς σε σχέση με τις εισαγωγές από τρίτες χώρες. Δεν θέλω να επενθυμίσω εδώ ότι είμαστε σε μια φάση συζητήσεων για αναθεωρημένο καθεστώς ε, φυτοϊγιεινής προστασίας το Κοινοβούλιο ε, τον Απρίλιο του 2014 στην Ολομερία του. Ε, ψήφισε. Ε, γίνανε λοιπόν συζητήσεις και συνεχίζονται συστήσεις με το Συμβούλιο. Τα κράτη-μέλη επιδιώκουν μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση σε σχέση με τα τρίτα κράτη και τις εξαγωγές, τους, εξαγωγές ε, μεγάλου, μεγάλου φάσματος φυτών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και σχετικούς περιορισμούς. Αντιλαμβάνομαι επίσης ότι σημείο εισόδου λέγεται πως ήταν το Ρότερνταμ. Δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτό, δηλαδή ότι ε, μπήκε μέσω του Ρότερνταμ αυτό το μικρόβιο. Όντως οι αρχές του Ρότερνταμ, ε, οι τελωνιακές, οι λιμανικές αρχές βρήκαν να εισάγονται πρόσφατα φυτά που έχουν νοσήσει, που νοσούν από την κλεψιέλα, αλλά δεν επιβεβαιώνεται ότι το πρώτο σημείο εισόδου, το αρχικό σημείο εισόδου ήταν εκλεψίελα. Αυτά και ελπίζω να έχω απαντήσει στις ερωτήσεις σας. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ο κύριος Μποβέ ζητάει το λόγο. Ναι, Πρόεδρε, και στο συγγνώμη που άργησα. Πάνω από μια μισή ώρα καθυστέρησε και το τρένο μου. Δυστυχώς μόνο τώρα μπορούσα να φτάσω. Ε, το Νοέμβριο απέστειλα ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μου, στην οποία μου απάντησε και γραπτός ε, η Επιτροπή για την κλεψιέλα. Αλλά το πρόβλημα επιδεινώνεται και στη Γαλλία, κυρίως στην Κορσική, επιδεινώνεται διότι είναι ξεκάθαρο ότι στην Κορσική έχουν εντοπιστεί δέντρα σε ε, καταστήματα που πολλούν σούπερ μάρκετ και το καθεξής, διακοσμητικά, φυτά, ελιάς, ελαιόδεντρα, τα οποία έχουν ε, εμφανεί τα σημάδια της κλεψίαλα. Γιατί λοιπόν δεν αναλαμβάνονται μέτρα. Πρέπει να λεφθούν μέτρα πολύ πιο αποτελεσματικά, να παρεμποδιστεί η κυκλοφορία αυτών των ελαιοδέντρων. Όπως η Αυστραλία παραδείγματι που εμποδίζει την είσοδο ιουδήποτε φυτού. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα να απαγορεύσει την είσοδο ιουδήποτε φυτού που μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την Ευρώπη. Δάλλως οδεύουμε προς την καταστροφή. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι δύσκολη κατάσταση. Και για τις διάφορες περιοχές και για τα είδη των φυτών στα οποία θα πρέπει να ενσκύψουν οι ερευνητές, η Επιτροπή να ενημερωθεί και να ενημερώσει και εμάς για τα μέτρα. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να διαδοθεί περισσότερο αυτή η ασθένεια. Και πρέπει να κοιτάξουμε πολύ προσεκτικά πώς ετέθησε η κυκλοφορία φυτό με την ασθένεια αυτή. Όλα αυτά πράγμα. πράγματα. Νομίζω ότι συζητήσαμε όσο μπορούσαμε το θέμα. Όπως είπαμε θα επανέλθουμε. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Αλλά τώρα δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο οπότε να το κλείσω και να περάσω στο σημείο 6. Τα κτηνιατρικά φάρμακα. Που θα συζητηθεί μαζί με το επόμενο θέμα, το υπαριθμό 7 με μια παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Αντζέρης είχε κάνει την παρουσίαση, τώρα θα γίνει συζήτηση. Αρμόδια κατ' ουσίαν περιβάλλοντος, εμείς έχουμε γνωμοδότηση. Ας ακούσουμε όμως, ας προχωρήσουμε τώρα, έχουμε ακούσει τον διευθυντή. Προτείνω να δούμε αν υπάρχουν ερωτήσεις ή παρατηρήσεις από τους συναδέλφους και μετά. Θα παρακαλέσω τους συντάκτες ε, των γνωμοδοτήσεων. Οι συνάδελφοι λοιπόν τώρα. Ερωτήσεις, παρατηρήσεις και η κυρία Πόλσιν και εσείς αν έχετε κάτι. Θέλετε να λάβετε το λόγο πρώτη, περιμένετε μετά, τώρα. Παρακαλώ λοιπόν, κύριε Πόλση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι συνοπτικότατη. Για το Ευρωκοινοβούλιο ήταν προφανές ε, το ψήφισμα εγκρίθηκε από την Επιτροπή Γεωργίας το 2011 και εκεί υπογραμμίσαμε την ανάγκη να διατηρηθεί η δραστικότητα των κτηνιατρικών φαρμάκων, ιδίω των αντιβιωτικών. Επίσης, ε, αναφερθήκαμε στην ε, φέβρεση νέων φαρμάκων. Γι' αυτό θελήσαμε να ορίσουμε και τον αγώνα κατά της μικροβιακής, μικροβιολογικής αντίστασης. Είναι μεγάλη μας ε, χαρά να διαβάζουμε τώρα ποιες είναι οι απόψεις του Κοινοβουλίου σχετικά. Απλώς δεν βλέπουμε να μεταφράζονται σε ένα πρόγραμμα πρωτοβουλειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της μικροβιακής αντίστασης. Στην ε, σημερινή μορφή της πρότασης, στο άρθρο 54, βρίσκουμε κάποια στοιχεία, όμως η πρόταση αυτή κανονισμού για τα κτηνιατρικά φάρμακα είναι απλώς ένα βηματάκι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ένα πολύ μικρό βήμα. Η όλη πρόταση είναι, πώς να το πω, κάπως ε, ε πολύπλοκη. Είναι δύσκολο να την καταλάβει κανείς. Είναι δυσνόητη και είναι και ε, αρκετά περίπλοκη. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναγνωρίσω ότι ένα πλεονέκτημα το έχει. θέλει να αντιμετωπίσει το γραφειοκρατικό άχθος. Όμως νομίζω ότι πράγματι η πρόταση αυτή θα πρέπει να απλουστευτεί έτσι ώστε ο όλος τομέας να έχει μια ευκαιρία να ανταγωνιστεί ισότιμα, ώστε η έρευνα, καινοτομία και η παραγωγή νέων φαρμάκων να ενθαρρυνθούν. Είναι σημαντικό τα κτηνιατρικά φάρμακα να είναι λιγότερο κερδοφόρα από ότι τα ανθρώπινα. Το πρόβλημα είναι κύριε Πρόεδρε ότι τα ζώα έχουν πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά. Γι' αυτό δεν υπάρχει αρκετή έρευνα. Δεν ε, φέρνει κέρδος αυτό για τους ερευνητές, γι' αυτό δεν εφευρίσκονται νέα φάρμακα. Ε, να κάνω εδώ κάποια σχόλια. Στο άρθρο 120 καταλαβαίνω ότι θέλουμε να περιορίσουμε την χρήση την ιατρικών φαρμάκων. Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να φροντίσουμε να απαγορευτεί η συνταγογράφηση από τους κτηνιάτρους. Ε, οι κτηνίατροι πρέπει να έχουν τις ίδιες αρμοδιότητες με τους γιατρούς ε, στους ανθρώπους. Όμως ορισμένα κράτη-μέλη, οι κτηνίατροι, έχουν γίνει απλώς συνταγογράφοι. Δεν είναι πλέον γιατροί των ζώων. Ενώ οι γιατροί ε, που ασχολούνται με τους ανθρώπους παίρνουν καλές αμοιβέ. Αυτό δεν ισχύει για τους κτηνιάτρους, γι' αυτό έχουν γίνει ακριβώς ε, συνταγογράφοι. Πρέπει λοιπόν να ορίσουμε πολύ σαφέστερα κριτήρια. Δεν μπορεί να είναι απλώς συνταγογράφοι, αλλά να κερδίζουν τη ζωή τους με τις ε, υπηρεσίες που προσφέρουν, όχι με τις συνταγές τους. Επίση, σε αυτή την νομοθετική πρόταση, Πρόεδρε, δεν υπάρχουν αρκετοί ορισμοί. Όταν θα φτάσουμε στο στάδιο των τροπολογιών βέβαια, θα μπορέσουμε να αναφερθούμε και στο πρόβλημα των ορισμών, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να απλουστευτεί η νομοθεσία. Νομίζω ότι αν καταφέρουμε να την απλουστεύσουμε, θα μπορέσουμε να είμαστε και ακριβέστεροι και σταθερότεροι και απλούστεροι στη χρήση ή της καταχρήσης των αντιβιωτικών. Σας ευχαριστώ. Ε, ούτως ή άλλως, συζήτηση θα γίνει στις 16 Απριλίου. Ε, περισσότερο λεπτομέρειες από τη σημερινή μας συνεδρίαση σήμερα. Θέλω απλώς να έχουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψε να δώσω τον λόγο και στον συνάδελφο Πόλτσακ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, πρέπει να πω ότι Για την ώρα δεν έχουμε μετάφραση. Αυτός είναι ο κανονισμός που προβλέπει τις διαδικασίες για την έγκριση και αδειοδότηση κτηνιατρικών φαρμάκων για κτηνιατρική και ανθρώπινη κατανάλωση για τα σχόλια της συναδέλφου Πάουλσεν για την χρήση κτηνιατρικών φαρμάκων και τη διαφορά τους με τα φάρμακα για ανθρώπους. Εγώ είμαι υπεύθυνος για το δεύτερο κομμάτι, που είμαι και συντάκτης της ε, γνωμοδότησης. Η Επιτροπή μας καλέθεται να καταγράψει τα εξής. Οι προτινόμενες αλλαγές για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρμοδιότητες της βάσης της συνθήκης της Λισαβόνας, ιδίως με τη διαδικασία της επιτροπολογίας που τώρα έχει αλλάξει από τη συνθήκη της Λισαβόνας, προβλέπει και αλλαγές που δεν έχουν σχέση με τον νέο κανονισμό για τα κτηνιατρικά φάρμακα και τη συνθήκη της Λισαβόνας. Χωρίς λοιπόν την απαραίτητη αξιολόγηση αντικτύπου δεν δικαιολογείται το πεδίο του κανονισμού καθώς και σε κάποια άλλα τμήματα της πρότασης. Αυτό αφορά κυρίως την κατάργηση των εξουσιών του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά τα τέλη που επιβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για την αδειοδότηση και την ε, καταγραφή και άλλων υπηρεσιών που ε, παριθμώντας τα ανάλογα άρθρα του κανονισμού αναφέρεται στο άρθρο 70 όπου λέγεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ορίσει τα τέλη ε, με εφαρμοστική πράξη. Θεωρώ ότι αυτό είναι τελείως άσκοπο ε, και μη ε, εύστοχο. Πολλά έχουν αναφέρει ότι ε, του ανησυχεί η μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Συμβούλιο προ την Επιτροπή. Όμω δεν είναι απλώ μια τεχνική τροπολογία. Έχει να κάνει με τι εξουσίε ε, και τη μεταφορά εξουσιών ε, εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Φαρμάκων προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο άρθρο 140 ο νέο κανονισμό δίνει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων νέε αρμοδιότητε για την μετάδοση πληροφοριών σε ό,τι αφορά τα μέλη τη Επιτροπή νομοποίηση των κτηνιατρικών φαρμάκων που προτείνονται από τα κράτη-μέλη. Εάν έπρεπε να συνοψίσω την ε, συνεισφορά μου εδώ ο κανονισμός που ορίζει την ε, ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και καθορίζει τις αρμοδιότητές του ε, προβλέπει και τη χρηματοδότηση των διαστηριοτήτων του, δηλαδή τον προπολογισμό του. Θεωρώ ότι αυτό μπορεί να γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευση, μπορεί να συζητηθεί περαιτέρω, αλλά κατά την άποψή μου απαιτεί μεγάλε αλλαγέ. Μπορώ να το συζητήσω με τους ε, συναδέλφους και όδου εισηγητέ, αλλά η βασική μου αντίρρηση έχει να κάνει με το άρθρο 70. Είναι το πιο προβληματικό σημείο. Ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλοι επτά που έχουν ζητήσει το λόγο, παρακαλώ έχει πάνω από ένα λεπτό ο καθένας. Στις 7 Απριλίου θα γίνει μια πλήρης αναπτυγμένη συζήτηση. Παρακαλώ ε, κρατηθείτε. Ρόσλινγκ. Ένα λεπτό είπαμε. Ναι, πολύ σύντομα. Γιατί λαμβάνονται τόσο λίγο υπόψη στην πρόταση επιτροπή τα εναλλακτικά μέσα και γιατί η μεταφυλακτική δεν αξιολογείται ως πρόβλημα. Γιατί είπα και νωρίτερα ότι τα δύο τρίτα των αντιβιωτικών που χρησιμοποιούνται χρησιμοποιούνται στην κτηνοτροφία. Ασφαλώς και πρέπει να περιοριστούν αυτά, γιατί δεν υπάρχει λοιπόν σχέδιο για μείωση, γιατί δεν ασχολείται η συζήτηση εκτός της άδεια και επιτάχυση των αδειών για τα αντιβιωτικά με τον περιορισμό της χρήσης. Ευχαριστώ πολύ σύντομα. Ναι, Πρόεδρε, μια πολύ συγκεκριμένη και τεχνικού τύπου ερώτηση, λέει ο κύριος Άγνιου. Συζητούμε τον κανονισμό για τα κτηνιατρικά ή για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση. Θα μας εξηγήσει λίγο, κυρία Πόλσεν, που βρισκόμαστε. Παρακαλώ. λέει. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα απαντήσω. Στις ερωτήσεις, Πρόεδρε, εγώ νομίζω ότι δεν χρειάζεται τώρα να ανοίξουμε πολύ τη συζήτηση του Άλλωστε θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τα θέματα αργότερα. Αυτό που θέλουμε όμως εδώ είναι να έχουμε, να αποφύγουμε μάλλον την αντιβιωτική προφύλαξη. Θέλουμε να περάσουμε στη χρήση μόνο σε περίπτωση θεραπείας και όχι προληπτικά των αντιβιωτικών. Αυτό όμως είναι το πιο σημαντικό. Πάμε Καπουτό. Κύριος Καπούτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επειδή θα συζητήσουμε και στις 16 Απριλίου, θα είμαι συνοπτικός. Να επισημάνω κάτι που είχα πει και άλλες φορές για τους ενδιασμούς μας. σε ό,τι αφορά τα κτηνιατρικά φάρμακα και τα φάρμακα για τους ανθρώπους, πέραν αυτών που υπόθηκαν προηγουμένως, και την αντιμικροβιακή αντίσταση, Πρέπει να ορίσουμε καλύτερε διαδικασίε αδειοδότηση και έγκριση. Πρέπει να προστεθούν και να είναι ενιαίε. Το ίδιο και η περίοδο προστασία και τήρηση των αρχείων τη τεχνική τεκμηρίωση μέχρι 18 χρόνια για να αποφύγουμε και τι δεσπόζουστε θέσει στην αγορά. Και για την επισήμανση. Τα λέω τώρα όσο πιο γρήγορα μπορώ τηλεγραφικά. Επτά κατηγορίε πληροφοριών προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμεί για λόγου διαφάνειας θέλουμε περισσότερε. Και για λόγου καλή γνώσης για του καταναλωτέ. Χρειάζονται πρόσθετε πληροφορίε. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί και στην ε, πώληση στο διαδίκτυο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δεύτερο σημείο που είναι και το τελευταίο για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, θεωρώ ότι σωστό είναι η διαδιδότηση να γίνεται από τον ίδιο οργανισμό που ασχολείται με τα ανθρώπινα φάρμακα, αλλά θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ η λειτουργία του στο δυνατόν συντομότερα. Ευχαριστώ. Κύριο Σταραμπέλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, πολύ γρήγορα εν ώψη της 16ης Απριλίου για την αντιμικροβιακή αντίσταση. Μία διάσταση του θέματος είναι, και ξέρω τη στάση της κυρία που είναι θετική, είναι να επιτρέψουμε στους κτηνιάτρους τη χορήγηση φαρμάκων. Διότι η διάγνωση πολλές φορές υποχρεώνει να χορηγηθεί το φαρμάκο στο δυνατόν πιο γρήγορα για να είναι δραστικό και αποτελεσματικό. Στον χώρο της κτηνοτροφίας αν αποσυνδέσουμε τη συνταγογράφηση από τη χορήγηση, ε, θα περάσει χρόνος ε, και θα μπορέσει να εξαπλωθεί γρήγορα η επιδημία σε πολλά ζώα του ζωικού κεφαλαίου, πράγματι κίνδυνο. Άρα όσο πιο γρήγορα μπορέσει ο κτηνίατρος να συνταγογραφήσει, τόσο το καλύτερο. Ξέρει τη δουλειά του και καλό είναι να μπορεί να χορηγήσει και το φάρμακο. Επίσης, το είπε και ο κύριος Ανδριουκάητης για την ε, ε, για τις οτροφές. Δουλειά των ε, κτηνιάτρων δεν είναι βεβαίως συνταγογράφηση, αλλά πρέπει να δούμε την αντιμικροβιακή αντίσταση και είναι καθοριστικό το πώς ε, τρέφουμε τα βοηδή, το ζωικοκεφάλαιο, τα πολερικά. Πρέπει αυτόν τον αγώνα της αντιμικροβιακής αντίστασης να τον πάμε μέχρι τέλους. Ευχαριστούμε η κυρία Αγκουλιέρα Γκαρσία. Eh, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω ότι συμφωνώ με αυτό το οποίο είπατε. Και αυτό που είπε η κυρία Πάουλσεν. Νομίζω ότι είναι περίεργο να απολύει τα φάρμακα για τα ζώα ο ίδιος ο κτηνίατρος. Για την κυρία Πάουλσεν τώρα, θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας για τον ορισμό της προφύλαξης, της μεταφύλαξης σε εισαγωγικά και το τι προβλέπει ο κανονισμός για τα κτηνιατρικά φάρμακα πέρα από τους τρόπους χορήγησης ε, των φαρμάκων Θα ήθελα την άποψή σας. Πρόεδρε, ένα δευτερόλεπτο ακόμα. Αυτό το οποίο είναι δύσκολο είναι ότι υπάρχουν διαφορετικές ε, μορφές χορήγησης και διαφορετικές μορφές αντίληψης της διαδικασίας χορήγησης. Αν ε, αποφασίσουμε μία μορφή τότε θα πρέπει να την κάνουμε σεβαστή και να υπάρχουν συγκεκριμένα όρια. Ευχαριστώ πολύ. Καταλαβαίνω ότι οι εισηγητές μας, ε, οι εισηγητές προς γνωμοδότηση έχουν όλοι σημειώσει τις επιφυλάξεις σας, το έκανε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν το θέλει της δίνω το λόγο για δύο με τρία λεπτά το πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα λίγα λόγια να μπορέσω να πω για την γνωμοδότηση ε, της ε, κυρίας Πάουλσεν. Είναι σαφές, ε, λέει ο εκπρόσωπος της Επιτροπής των Περιφερειών, ότι θα πρέπει να πλουστεύσουμε τις διαδικασίες αδειοδότησης και να δώσουμε κίνητρα για την καινοτομία αυτό είναι κάτι το δύσκολο. Ε, σαν παράδειγμα η προστασία των ευρεσιτεχνιών, η διάρκεια τους ε, είναι ικανοποιητική για τους ε, κτηνιάτρους και για τους ε, εμπόρους των φαρμάκων αυτών. Μήπως θα πρέπει να υπάρξει μια μεγαλύτερη χρονική περίοδος κάλυψης. Ταυτόχρονα θα ήθελα να υπάρχουν κοινέ ευθύνε εδώ και όχι με μονομένα ημίμετρα. Ευχαριστώ. Ε, για δύο-τρία λεπτά ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την κυρία Πάουλσεν και όλους που πήραν μέρος σε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να πω σύντομα ότι προσπαθούμε να μειώσουμε τα, την γραφειοκρατία και θα σας παρουσιάσουμε τα μέτρα αυτά στην επόμενη αναλυτική συζήτηση. Είναι αλήθεια ότι η πρόταση είναι μια περίπλοκη πρόταση, διότι καλούμεθα να κωδικοποιήσουμε όλες τις νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες καλούνται να διαχειριστούν το θέμα αυτό το τόσο σημαντικό για την υγεία των ζώων αλλά και για την υγεία γενικότερα. Έχουμε διευρύνει το χρόνο προστασίας των ε, ε, συγκεκριμένων στοιχείων που επιτρέπει σε ε, αυτούς που ασχολούνται με την καινοτομία να εφεύρουν, να δημιουργήσουν νέου τύπου φάρμακα. Έχουμε ασχοληθεί και με το θέμα της χορήγησης και της συνταγογράφησης των φαρμάκων. Από τη μία θα πρέπει εμείς να πάρουμε τις σωστές πρωτοβουλίες για τους επαγγελματίες. Από την άλλη θα πρέπει να μην αγνοήσουμε ε, το ευρύτερο πρόβλημα που, έχουμε, που καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε ιδιαίτερα σε ορισμένες χώρες ε, της καταπολέμησης της αντίστασης στα αντιβιωτικά. της αντίστασης ε, στα μικρόβια περισσότερο. Λοιπόν, ε, σχετικά τώρα με την τελευταία παρατήρηση να αναφερθώ σε μία απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου το οποίο ουσιαστικά δημιουργεί νομολογία, συστήνει αν θέλετε, ε, την περίπτωση της ε, εξωτερικής υπηρεσίας για τα χημικά, ότι θα πρέπει δηλαδή να υπάρξει μια αντίστοιχη ρύθμιση και για τα φάρμακα, αποδίδοντας ε, ουσιαστικά τον πλήρη έλεγχο στο Συμβούλιο. Έχουμε επίσης ε, θέσει και το θέμα των τελών για την προφύλαξη το από φαρμακευτικές ουσίες. Υπάρχει πρόβλημα για τις παραγγελίες ε, διαδικτυακά φαρμακευτικών ουσιών. Εμείς πιστεύουμε όμως ότι μια καλή ε, καλώς ρυθμιζόμενη παραγγελία φαρμάκων διαδικτυακά να βοηθήσει να φτάσουν οι ουσίες αυτές σε συγκεκριμένες περιοχές. Αυτό όμως θα πρέπει να γίνεται με τον σωστό έλεγχο. Και όλα τα, όλα τα τμήματα, τα επιμέρους τμήματα του συστήματος θα πρέπει να ρυθμίζονται σωστά. Για την αντίσταση τώρα στα μικρόβια, Έχουμε το πρόγραμμα δράσης σε 12 σημεία, το οποίο εφαρμόζει στην παρούσα φάση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμμετέχει η ΕΦΣΑ, η EMA και η CD. It's an action plan, but, number of measures, uh, including this new regulatory framework. We... Και το νέο ε, ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο προτείνουμε νομίζω ότι έχει αρκετά μεγάλη σημασία για να μπορέσουν να συνεργαστούν σωστά γιατί αν δεν συνδυάσουμε το κτηνιατρικό κομμάτι, την φροντίδα των ζώων και την φροντίδα των ανθρώπων, από την άλλη με τα δίκτυα που παρέχουν τις φαρμακευτικές ουσίες, δεν θα καλύψουμε όλες τις πλευρές. Πώς θα λειτουργήσουμε λοιπόν προφυλακτικά, πώς θα ελέγξουμε τις συνέπειες μετά την χορήγηση των φαρμακευτικών ουσιών, Όλα αυτά μπορεί να τα δει η Επιτροπή ε, η Ευρωπαϊκή για τα φάρμακα που ασχολείται ειδικότερα με το θέμα. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε όλους τους ε, εκπροσώπους της Επιτροπής. Όπως σας το είπα θα το ξαναδούμε το θέμα στις 16 Απριλίου. Μπορείτε να υποβάλλετε τις τροπολογίες σας ως τις 24 του Απρίλη, οπότε έχουμε και άλλο χρόνο για να προετοιμαστούμε. Μιλώ για τα δύο σχέδια γνωμοδότησης. Και μπορείτε να θέσετε τις ερωτήσεις σας απευθείας στην Επιτροπή. Περνάμε τώρα στο σημείο 8 για την υγεία των ζώων. Η συγγήτρια η κυρία Πάουλσεν πάλι. Κυρία Πάουλσεν, ξέρουμε ότι ο τομέας αυτός παρουσιάζει ιδιαίτερη κινητικότητα. Ξέρουμε και τι κάνετε, υπάρχουν συστηματικά τριμερείς διάλογοι. Θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε εντάχει για τις πρόσφατες εξελίξεις. Και να μας πείτε που έχουμε φτάσει σήμερα στις συζητήσεις. Σας ευχαριστούμε και πάλι και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχουμε προχωρήσει αρκετά. Ήμουν εισηγητρία αρκετών νομοθετημάτων πολύ σημαντικών ναι, για αρκετά χρόνια. Τα θέματα αυτά ναι. πολλά ζητήματα πρέπει να εξετάσουμε προσοχή. Έχουν λοιπόν συνεργαστεί τα τρία θεσμικά όργανα με το προσωπικό τους. Και είναι πολύ ενδιαφέρον κύριε Πρόεδρε, διότι οι προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πέρασαν σε πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Μπορέσαμε δηλαδή να εξασφαλίσουμε την έγκριση των θέσεών μας. Τρεις τριμερείς διαλόγους με τελευταίο αυτόν της 13ης Μαρτίου διεξαγάγαμε Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε έτσι να ολοκληρώσουμε και να κλείσουμε με έναν τέταρτο τριμερή διάλογο που θα μας επιτρέψει να καταλήξουμε στα πιο απτά αποτελέσματα. Παραμένουν βέβαια εκκρεμή τα ζητήματα τα σχετικά με τις εκτελεστικές και τις κατεξουσιοδότησης πράξεις που είναι σημαντικές. Θα έλεγα ότι κάπου έχουμε συγκρούσεις, δεν μπορώ να το αρνηθώ κύριε Πρόεδρε, σε ορισμένα σημεία, αλλά πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να ε, καταλήξουμε σε μια συμφωνία και θα επανέλθω για να σας ενημερώσω όταν είναι όριμο το θέμα, όταν θα έχουμε κάποια λύση. Αλλά ήθελα να πω εξ αρχής ότι βρισκόμαστε ήδη στο σωστό δρόμο. Και ελπίζω την άλλη φορά να έχουμε και πιο πολύ χρόνο να το συστήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Πολύ καλά. Και σας ευχόμαστε πολλές επιτυχίες και στο μέλλον ώστε να γίνουν σεβαστές και οι προθεσμίες που έχουμε. Εάν οι συναδελφοί έχουν ερωτήσεις, παρακαλώ, αλλά δεν ενθαρρύνω. Δεν βλέπω να ζητάει κανείς στο λόγο λοιπόν. Καλώ, σας ευχαριστώ για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε. Ολοκληρώνουμε έτσι το σημείο αυτό της συνεδρίασης και προχωρούμε στους συντονιστέ μας για τους λοιπούς 9 το πρωί αύριο ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο. Και σας καλώ να είστε όλοι στην ώρα σας στην αίθουσα ώστε να μην χρειαστεί να περιμένει ο Επίτροπος 10-15 λεπτά μέχρι να γεμίσει η αίθουσα. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και ψηφοφορίες. Μία ψηφοφορία για την ψηφοφορία. Φαντάζομαι ότι αρκετοί θα έρθουν σε 9 ακριβώς για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ. Συντονιστές, συνεργάτες τους, και οι λοιποί αποχωρούν αύριο με τον Επίτροπο Χόγκαν.